Um, Καλησπέρα σας συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας συνεδρίαση. Ε, έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. σημειώσετε ότι δυστυχώς δεν θα έχουμε μετάφραση στα μαλτέζικα, στα ιρλανδέζικα και και στα κροατικά. Ε, τώρα βλέπουμε εδώ έχουμε μια έκθεση φωτογραφίας ε, στην επέτειο της πενταετίας της ΕΑΖΟ και θα γίνει μια παρουσίαση από τον κύριο Νίντελ Μίλερ για την ΕΑΖΟ και θα έχουμε και μια προβολή ταυτόχρονα για την επέτειο των πέντε ετών από την ε, δημιουργία της ΕΑΖΟ και ευχαριστούμε τους συναδέλφους που ε, κάνουν τη σημερινή έκθεση. Αυτά λοιπόν επεξηγηματικά για να καταλάβετε τι είναι αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε στην αίθουσα σήμερα. Τώρα, να εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών υπό τον κανονισμό 205 έχουμε τον ορισμό των εισηγητών καταρχάς για τον πρόεδρο υπό την κανόνα 50 της απλοποιημένης διαδικασίας έχουμε αυτοματοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων όσον αφορά στοιχεία DNA με τη Δανία και επίσης για τα δακτυλοσκοπικά στοιχεία πάλι στη Δανία σύμφωνα πάντα με το άρθρο 50. Η κυρία Γκάμπριλ του ΕΛΚ έχει οριστεί η συγγήτρια για την συμφωνία για επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Europol. Για γνωμοδότηση έχει οριστεί η κυρία Μάκο Βέη, η συγγήτρια, για την ε, κινητοποίηση του περιθωρίου που προβλέπεται για το 2017 2016 από την Επιτροπή Προϋπολογισμού και ζητώ, ρωτώ, σας ρωτώ αν εγκρίνετε αυτές τις συστάσεις των συντονιστών. Επίσης μια υπενθύμηση συνάδελφοι, ε, την κάρτα ψηφοφορίας σας να έχετε, γιατί θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες στις 5 και 40, 17 και 40. Περνάμε τώρα στο σημείο 3 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Ζήλ Ντεκερκόφ που είναι ο Ευρωπαίος Συντονιστής ε, της Αντιτρομοκρατικής ε, ευρωπαϊκής προσπάθειας μετά από τις πρόσφατες επιθέσεις στα κράτη-μέλη. Θα θυμάστε ότι στις 31 Αυγούστου είχαμε μία συζήτηση με την Προεδρία του Συμβουλίου για τις πρόσφατες αυτές επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις και τότε είπαμε ότι ο κύριος Ντεκερκόφ δεν είχε μπορέσει να έρθει αλλά θα εξασφαλίζαμε την παρουσία του εδώ ε, ενώπιόν μας στην ε, πιο σύντομη ε, δυνατότητα που υπήρχε και γι' αυτό και με χαρά το καλωσορίζουμε σήμερα εδώ ώστε να ενημερωθούμε για την κατάσταση ασφαλείας και να του θέσουμε τις ερωτήσεις που επιθυμούμε. Βεβαίω από τότε που τελευταία φορά τον είδαμε στην Επιτροπή μας και από τότε που είχαμε αυτή την ε, συζήτηση είχαμε και τις ακροάσεις ε, με τον Επίτροπο για την Ασφάλεια. Σίγουρα λοιπόν θα μπορούσε να μας πει και δύο λόγια για το πώς θα συνεργαστεί με τον Επίτροπο για την Ασφάλεια, πώς θα επηρεαστεί και πώς θα γίνει μάλλον συντονισμό σε αυτό το τομέα και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεκέρκοφ. Και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Αυτό το λόγο κύριε Τεκερκόφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ καταρχήν που με καλέσατε. Δεν μπόρεσα να είμαι παρόν στο τέλος του καλοκαιριού στην πρώτη συζήτηση που είχατε για το θέμα αυτό και θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στα διδάγματα από τις πρόσφατες επιθέσεις και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε υπό το φως αυτών των ε, διδαγμάτων. Αρχές Σεπτεμβρίου ήμουν ε, με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών, τον Καζνεύ, και μιλήσαμε για τον κίνδυνο και τις απειλές που είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, το υψηλότερο τα τελευταία 20 χρόνια. Και αυτό κυρίως διότι οι απειλές αυτές ε, έχουν πολύ διαφορετικές ε, αιτίες και μορφές. Έξι χαρακτηριστικά μπορούμε να εντοπίσουμε. Πρώτον, πολλά διαφορετικά προφίλ δραστών. Δίκτυα, ομάδες, τζιχαντιστές που στέλνονται από τη Ράκα, Εκεί υπάρχει μια μονάδα σχεδιασμού επιθέσεων και ακόμα και αν οι επικεφαλείς έχουν δολοφονηθεί, παρόλα αυτά συνεχίζει ο σχεδιασμός των επιθέσεων. Επίσης έχουμε και τους ε, μοναχικούς ε, δράστες, μαχητές, οι οποίοι δεν δρούν τόσο πολύ μοναχικά, διότι από κάπου εμπνέονται. Υπάρχει ο περίφημος Γάλλος ε, καθοδηγητής ο Ρασίμ Κασίμ, ο Ρασίτ Κασίμ, ο οποίος ε, χρησιμοποιεί το σύστημα Telegram για να κατευθύνει τις επιθέσεις. Πρόκειται δηλαδή για άτομα τα οποία εμπνέονται από τα μήνυματά του, από την προπαγάνδα του. Και η τρίτη κατηγορία είναι τις περισσότερες φορές άτομα ψυχοπαθή ή που ψάχνουν ε, να αυτοεπιβεβαιωθούν ή να μιμηθούν ε, γεγονότα που έχουν συμβεί με άλλους. Δυστυχώς ο κεντρικός ρόλος του διαδικτύου αυτή τη στιγμή είναι η διάδοση αυτών των ιδεών, αυτής της ιδεολογίας, αλλά η καθοδήγηση με κωδικοποιημένα μηνύματα τέτοιων επιθέσεων. Είναι κάτι το οποίο ακόμα και αν δεν μας αρέσει θα πρέπει σαφώς να το παραδεχτούμε ότι χρησιμοποιούνται τα μεταναστευτικά ρεύματα, η πλαστογράφηση εγγράφων, για να ενσωματωθούν κάποιοι μέσα σε αυτές τις ροές, κάποιοι τρομοκράτες. Στην Ευρώπη έχουμε ανιχνεύσει, έχουμε εντοπίσει, δεν μπορώ να σας δώσω πολύ συγκεκριμένους αριθμούς, εκατοντάδες πάντως τέτοιους δράστες οι οποίοι έχουν εγκληματικό παρελθόν, έχουν δηλαδή ποινικό μητρό, είτε χρησιμοποιούν αυτό το οργανωμένο έγκλημα για να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατική τους δράση. Και αυτό έχει τις εξής συνέπειες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να εντοπίσουμε εγκαίρως την ριζοσπαστικοποίηση. Δηλαδή πολλές φορές ψάχνουμε κάποιον ο οποίος έχει μια συμπεριφορά ή τουλάχιστον δεν συμπεριφέρεται όπως ε, θα περιμέναμε να συμπεριφέρεται κάποιος ο οποίος διακατέχεται από την ιδεολογία του τζιχάντ. Δεύτερον, πολλές φορές βλέπουμε άτομα τα οποία προσπαθούν να βρουν πλαστά έγγραφα, εξοπλισμό και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να βρουν χρηματοδότηση για να φτάσουν μέχρι αυτό τον εξοπλισμό. Τρίτο, πώ οργανώνονται αυτές οι επιθέσεις και ποιο είναι το modus operandi. Είδαμε παραδείγματος χάρη στο Παρίσι, στο Μπατακλάν, υπήρχε πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Άλλε φορές βλέπουμε πιο μεγάλο αυτοσχεδιασμό. Είναι κάτι που βεβαίως ε, μας οδηγεί σε μια διαφορετική ανάλυση αυτών των γεγονότων που δεν είναι πλέον ε, συμβολικές. Υπήρξαν επίσης και επιθέσεις σε μουσουλμανικές χώρες με αποτέλεσμα να αποτρέψουν τον τουρισμό σε χώρες όπως η Τινησία, η Αίγυπτος και η Τουρκία που ε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και από τα έσοδα του τουρισμού και τέλος, αυτό που θα ήθελα επίσης να προσθέσω είναι ότι όταν ε, παρακολουθεί κανείς τις επικοινωνίες διαπιστώνει ότι υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα. Οι επιθέσεις ε, του ΝΤΕΣ πρόκειται να αλλάξουν μόντους οπεράντι, χρησιμοποίηση ε, κρυκτικά σε αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη, και βεβαίως η χρησιμοποίηση των ε, μαχητών οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες στην Ευρώπη ε, ο επαναπατρισμός. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι όταν καταρρεύσει το Καλυφάτο, το ISIS, όλοι αυτοί οι όχι εκατοντάδες αλλά χιλιάδες πλέον ε, μαχητές θα προσπαθήσουν είτε να κρυφτούν κάπου, όπως παραδείγματος χάρη στη Λιβύη, είτε να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Και θα έχουμε βεβαίως πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και κατηγορίες ε, μαχητών. Αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, όμως ε, κάποιοι οι οποίοι είναι εξίσου επικίνδυνοι και οι οποίοι βρίσκονται στις πίσω γραμμές, αλλά και πολλές ε, γυναίκες και παιδιά, πολλά παιδιά, πολλοί ανήλικοι μαχητές. Είδαμε σε πολλές χώρες, όπως παραδείγματο χάρη ε, τη Γερμανία, με πολλούς ε, πρόσφυγες, προσπάθεια να ενσωματωθούν στις ομάδες των σαλαφιστών παραδείγματος χάρη άτομα που βρίσκονται μεταξύ των προσφύγων. Και βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει και την Ισλαμοφωνία, τον φόβο ε, προς ε, το Ισλάμ και την ε, ριζοσπαστικοποίηση. Το θέμα της Λιβύης επίσης το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα, η Λιβύη η οποία μπορεί να δημιουργηθεί στην οποία μπορεί να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα από όπου θα ξεκινάνε όλες οι επιθέσεις του ΝΤΑΕΣ. Η οργάνωση Τζαπατά Αλνούστρα, παραδείγματο χάρη, η Αλκάιντα που σήμερα αντιμάχεται τον Ασάτ, που μπορεί όμως ε, να στοχεύσει και τη Δύση. Σε κάθε περίπτωση, κάποια από τα διδάγματα που θα πρέπει να αποκομίσουμε από τις πρόσφατες επιθέσεις είναι ότι σήμερα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την κινητοποίηση των ε, θεσμικών οργάνων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχει ένας επίτροπος αρμόδιος ε, για το θέμα αυτό, κάτι που σίγουρα θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα. Ακούσατε τις δηλώσεις του, η μία είναι για την πρόληψη και η άλλη για την ασφάλεια. Η Ένωση της Ασφάλειας είναι κάτι που παίρνει σάρκα και οστά και που σίγουρα θα ενδυναμώσει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εσωτερική ασφάλεια. Η δράση της Επιτροπής ε, είναι αποφασιστική και σκοπός μας είναι βεβαίως να βελτιώσουμε και τις ε, επαφές μας με τις ε, χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου. Ήμασταν πολύ πρόσφατα στην Ιορδανία, το Λίβανο, την Τινησία, την Αίγυπτο, Αλγερία με σκοπό να τους στηρίξουμε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό του είδους της δυσκολίας. Είδατε μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής της Μπρατισλάβα ότι το Συμβούλιο εκφράζει πλέον την αποφασιστικότητά του. Η αντιτρομοκρατική δράση βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Συμβουλίου η διαδικασία στην Πρατισλάβα έχει ξεκινήσει, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ε, νέες βάσεις δεδομένων που αφορούν την ριζοσπαστικοποίηση. Ποιες είναι οι προκλήσεις ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτη πρόκληση, συλλογή πληροφοριών, ενημέρωση, και ανάλυση των δεδομένων που διαθέτουμε. Εδώ πρέπει να γίνει βεβαίως πάρα πολλή δουλειά με τις δύο νέες βάσεις δεδομένων που προτείνει η Επιτροπή ΕΣΤΑ για αυτούς που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεωρήσεις και τις εξόδους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η διαδικασία στην απόφαση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει εδώ σύνδεση των δεδομένων μέσω αυτών των δύο βάσεων. Δεύτερον, αξιολόγηση της ε, συνισφοράς των ε, κρατών μελών προς αυτές τις δύο βάσεις δεδομένων. Όλα τα κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες έχουν ε, συνεισφέρει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο έχουν βελτιώσει τη συνεισφορά τους τα κράτη-μέλη. Δηλαδή το δίκτυο της Europol, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν τους ε, συνδέσμους τους που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο αυτό της Europol και χρησιμοποιούνται αυτές ε, οι βάσεις δεδομένων, αυτές οι δυνατότητες πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Το ISS καθώς και η επαγρύπνηση βάση του άρθρου 36. Αναφέρομαι εδώ στην δυνατότητα συναγερμού έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις συναγερμού κατά 400% μεταξύ 2004-2016. Σήμερα έχουμε πάνω από 9.000 ε, τέτοιου είδους ε, συναγερμούς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει και απαιτεί τη συνεισφορά όλων. Γνωρίζω βεβαίω ότι εδώ υπάρχουν και οι περιορισμοί βάσει της ε, αρχής της προστασίας των δεδομένων. Και βεβαίως εδώ η αρχή της, περιορισμένη περιορισμένης χρήσης των δεδομένων είναι κάτι το οποίο σαφώς θα πρέπει να διέπει αυτήν την δραστηριότητά μας. Αν θέλουμε όμως κάποιος που βρίσκεται στα σύνορα να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να μπορέσει να συνειδητοποιήσει μεταξύ των μεταναστών ποιοι είναι απλώς λαθρομετανάστες, ποιοι ζητούν άσυλο και ποιοι ε, πρόκειται να μπουν σε μια άλλη κατηγορία, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα δίκτυα με όλα τα βιομετρικά στοιχεία και σε κάθε περίπτωση η αρχή της προστασίας των δεδομένων εδώ θα πρέπει με κάποια ευελιξία να αντιμετωπιστεί. Η ομάδα υψηλού επίπεδου που έχει ήδη συναντηθεί δύο φορές συνεχίζει τις εργασίες της και είμαι πεπισμένος ότι η πολύ φιλόδοξη εργασία της θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιουνιό του 2017. Το τρίτο σημείο που ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί είναι να δημιουργηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός είδους γέφυρα μεταξύ αυτών που ε, έχει δημιουργήσει η Europol με το κέντρο αντιτρομοκρατικής δράσης και την πλατφόρμα των ε, υπηρεσιών ασφαλείας, της ομάδας δηλαδή αντιτρομοκρατικής δράσης. Αυτό δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι υπάρχουν ε, κάποιες δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα ότι το θέμα των ε, πληροφοριών, των υπηρεσιών πληροφοριών είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Θα πρέπει όμως να βρεθεί σε κάθε περίπτωση ένας τρόπος, ένας μηχανισμός έτσι ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορέσουν να αποκτήσουν διασυνδέσεις. Το θέμα τώρα της συλλογής δεδομένων και της ανταλλαγής δεδομένων. Η Επιτροπή εδώ εξετάζει όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσει την Επιτροπή αρμόδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα το θέμα επίσης των ψηφιακών ε, δεδομένων. Η Eurova, η Επίτροπος ε, στις συνομιλίες που είχε με τις Ηνωμένε Πολιτείες επανέλαβε την ανάγκη εδώ να υπάρξει μία άμεση και ε, υψηλής ταχύτητας επικοινωνία. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτές οι προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε πολύ πιο άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Η Το επόμενο είναι ότι στην Κομισιόν πρέπει να κάνουμε μαζικές επενδύσεις στην πρόληψη. Όπως είπαμε, έχουμε όλο ένα και λιγότερους Ευρωπαίους που πηγαίνουν στη Συρία, γιατί είναι δυσκολότερη πρόσβαση αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε περισσότερους οι οποίοι ε, ε, ε επιστρέφουν από τη Ράκα ή από αλλού. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερο στο ίντερνετ μέσω αυτού του φόρουμ που έχει φτιάξει η Κομισιόν ε, και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και μια δεύτερη συνάντηση με τις εταιρείες ίντερνετ. Ε, περιμένω πολλά από εκείνες. Η ταχύτητα με την οποία θα αφαιρέσουν ε, το παράνομο περιεχόμενο και μάλιστα η εξέβρεση ενός αυτοματοποιημένου τρόπου για να γίνεται αυτό είναι πολύ σημαντική, καθώς και η στήριξη που μπορεί να δώσουν οι εταιρείε αυτές στην κοινωνία των πολιτών ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη ε, αντίθετου, ε, όπως λέμε, περιεχομένου. Άλλη σημαντική πτυχή που μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά, αλλά αυτό είναι και στην ανακοίνωση του Επιτροπής, είναι πώς μπορούμε να βάλουμε αφήνουμε το πρόβλημα και σε διάφορα άλλα ε, ε, τομείς ε, παιδείας, πολιτισμού, πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης, στον αθλητισμό κτλ. Πώς δηλαδή θα μπορούσε να μπει αυτό το θέμα σε όλους τους τομείς, έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Θα πρέπει αυτό να, μην, να είναι βέβαια ξεχωριστό, να μην θεωρηθεί ότι είναι ο βασικός στόχος η αντιτρομοκρατική δράση, αλλά να εντάσσεται μέσα σε όλα τα, τις εκδηλώσεις. Και τέλος, αποκατάσταση. Ανέφερα ήδη προηγουμένως, παλιότερα μάλλον, ε, στην Επιτροπή ότι δεν προχωράμε σε αυτό το τομέα. Δεν προοδεύουμε. Εάν θέλουμε να έχουμε ε, μια εργαλειοθήκη με όλες τις απαραίτητες ε, ε, πολιτικές ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε, να χωνέψουμε αυτούς τους μαχητές, θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε και εναλλακτικέ στη φυλακή και στις διώξεις. Δεν έχω το χρόνο να αναφέρω τα σύνορα. Ξέρετε πολύ καλύτερα τη μεταμόρφωση του Frontex, την εργασία για τα πλαστά έγγραφα, του συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και αναμένουμε ταχεία ολοκλήρωση των αλλαγών του Σέγγεν γιατί είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθεί αυτή η νομοθεσία. Επίσης δεν χρειάζεται να επεκταθώ στο εξωτερικό κομμάτι, αλλά ευχαρίστω θα σας εξηγήσω ε, τι θέλουμε να επιτύχουμε με όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ. Σας έκοψα λίγο γιατί περιμένουμε ερωτήσεις λεπτομερείς από τους ε, συναδέλφους. αν δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως εκείνους. Μπάρμπαρα. Παρακαλώ, δύο λεπτά έκαστος. Μπάρμπαρα Καρτίκα, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, εισήγηση. Ήταν ε, πάρα πολύ περιεκτικά τα όσα είπατε. Βέβαια δεν είναι εύκολο ε, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, ιδιαίτερα στη σήμερα εποχή. Ναι, έχουμε την εντύπωση ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην, στον αγώνα ε, κατά της τρομοκρατίας θα ήταν ε, μια γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων όσο το δυνατόν πιο γρήγορο, διότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ούτω ώστε ε, να μπορούμε να δρούμε από κοινού όταν υπάρχει κίνδυνος επιθέσεων. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, όσον αφορά τη χρήση δεδομένων και την ανταλλαγή αυτών μεταξύ των κρατών μελών θα ήταν ίσως μια δυνατότητα να ε, τα βρίσκουμε αυτά από άλλους ε, πόρους. Ε, αναφέρεται ότι θα υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Τι λοιπόν αντιλαμβάνεστε εσύ, τι εννοείτε όταν λέτε αυτά, τα, αυτές τις άλλες πηγές. Καταλαβαίνω ότι όταν οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας ε, δεν μπορούν να βρουν τα συγκεκριμένα ε, δεδομένα και δεν θέλουν να τα ανταλλάξουν, τότε η κατάσταση είναι δύσκολη. Όμως δεν θα ήταν καλύτερο αν προσπαθούσαμε να επιτύχουμε μια καλύτερη συνεργασία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, ούτως ώστε να μην έχουμε τις ίδιες δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, που δεν ήρθα από την αρχή της συνεδρίασης. Όμως έχω κάποια ερωτήματα. Το ένα αφορά και πάλι το ζήτημα όταν μιλάμε για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και αυτή τη διάκριση τότε φαντάζομαι ότι ε, δεν ανταλλάζουμε άβουλα κάποιες πληροφορίες, αλλά υπάρχουν οι αποδείξεις ότι εδώ κάποιος είναι ε, επικίνδυνος. Ε, γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μου πείτε πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει στο ζήτημα των κοινών κριτηρίων για ποιον λόγο κάποιος στα διάφορα κράτη-μέλη μπορεί να μπει σε μια τέτοια λίστα επικίνδυνων προσώπων. Είναι κάτι συγκρίσιμο ή εδώ θα πρέπει για άλλη μια φορά να βελτιωθούμε. Το δεύτερο δεύτερο αφορά το ζήτημα των ε, ε, αλλοδαπών μαχητών και κατά πόσο χρησιμοποιούν ε, τις διαδρομές των προσφύγων για να φτάσουν στην Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι ο Άισις δεν έχει καμία όρεξη έναν εκπαιδευμένο μαχητή να το στείλει μέσω ενός αβέβαιου δρόμου, μέσω του Αιγαίου για παράδειγμα, ίσως ε, λογικά θα έχει άλλους δρόμους ε, για να τους φτάσει στην Ευρώπη. Έχετε λοιπόν ε, για αυτό πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται αυτό. Τρίτον, στο τέλος της ομιλίας σας αναφέρατε ότι όσον αφορά την πρόληψη δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και με άλλους παράγοντες μέσα στις κατατόπους κοινωνίες, η δική μου εντύπωση είναι ότι πολλοί από τους θύτες, σχεδόν όλοι τους, δεν έχουν έρθει σε εμάς ως υπηκοϊτροί των χωρών, αλλά έχουν ζήσει από, από παλαιότερα στην Ευρώπη και ήδη στο εσωτερικό της Ευρώπης έκαναν τα πρώτα βήματα προς την ριζοσπαστικοποίηση το ερώτημά μου λοιπόν είναι ότι ακούω συνεχώς ότι σε αυτό το τομέα θα πρέπει να συνεργαστούμε με κατατόπους παράγοντες και εκεί να προωθήσουμε την πρόληψη. Όμως η δική μου εντύπωση ή και εδώ θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση ότι θα έπρεπε ε, να αξιοποιήσουμε περισσότερο προσωπικά, ε, προσωπικό και χρήματα ε, για να κλείσουμε τα σύνορα, να δημιουργήσουμε μεγάλες βάσεις δεδομένων, όμως είμαστε πιο συγκρατημένοι στα ίδια τα κράτη-μέλη και να κάνουμε εκεί την αναγκαία πρόληψη. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό και έχετε στοιχεία πάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Μπριγκίτ. Πριν περάσουμε στον επόμενο μιλτή, θα ήθελα να πω, το αναφέραμε αυτό στις ανακοινώσεις, αλλά δεν είχατε έρθει ακόμα, ότι εδώ είναι η τελευταία συνάντηση του κυρίου Κύρκου και θα φύγει μετά από αυτήν. Και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα είναι η τελευταία του συνάντηση εδώ. Θα θέλαμε λοιπόν να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά του. Είναι ένα πολύ καλός φίλος και είναι ωραίο να βλέπεις μέλη τα οποία εργάζονται τόσο σκληρά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα λοιπόν. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ένας ε, πολιτικός υπέρ της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για το έργο σας σε αυτή την Επιτροπή. Okay, and now you can ask your Και τώρα μπορείτε να θέσετε το ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Η τελευταία μου ε, δουλειά σε αυτή την επιτροπή θα είναι να ψηφίσω. Θα είμαι λοιπόν και πάλι εδώ το απόγευμα για να ψηφίσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας ε, σχόλια. Βρίσκομαι εδώ για 17 χρόνια και ελπίζεις ότι όταν έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία πάνω στα όσα κάνεις τότε θα γίνεις καλύτερος ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο καλεσπένος μας έχει αυτή τη θητεία εδώ και 9 χρόνια, αν έχω καταλάβει καλά, και πιστεύω ότι οι ευθύνε που έχει και τα όσα κάνει έχουν γίνει όλο και πιο ε, σημαντικά καθώς ο χρόνος περνά. Τα 9 χρόνια εμπειρία είναι πολύ σημαντικά για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω δύο πράγματα. Το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συντονιστής λοιπόν αντιτομοκρατικής δράσης δεν έχει πολύ ε, εξουσία όμως, νομοθετική εξουσία και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι μέσω της Επιτροπής μας αλλά και του Κοινοβουλίου μας θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη ώστε ο ίδιος ε, να ε, έχει ένα μεγαλύτερο ρόλο στις αντιδρομοκρατικές δράσεις του Συμβουλίου. Πολλά από τα πράγματα που κάνει είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς το CTC θα συντονίσει το, ε, νέο, τη νέα υπηρεσία αντιτρομοκρατικής δράσης της Europol και χαίρομαι που ο νέος Επίτροπος ε, για την ε, Ασφάλεια της Ένωσης είναι Βρετανός και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω πώς βλέπει το δικό του ρόλο εργαζόμενος ε, σε συνεργασία με τον Σερ Τζούλιαν. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είχα μια πολύ ωραία εμπειρία εργαζόμενος σε αυτή την εμπειρία και ναι κύριε Πρόεδρε έχετε δίκιο ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου εδώ σωστά αν δεν μπορούσα αν δεν είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ με μέλη όλων των ε, πολιτικών ομάδων διότι πιστεύω ότι αυτό που, μπορούμε να, που προσπαθούμε να κάνουμε αφορά το κοινό καλό των Ευρωπαίων πολιτών και πιστεύω ότι η Επιτροπή αυτή θα μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει με πλήρη εκπροσώπηση και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Σισίλια τώρα. Ωραία. Θα δώσω το λόγο στη, ε, στη συνάδελφό μου Σόφη. Σόφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ στον κύριο Ντεκέρκοφε για την παρουσίαση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Ε, μαζί με αυτά που είπε ο Τίμωθη. Χαίρομαι ιδιαίτερως που δημιουργήθηκε ένα καινούριο χαρτοφυλάκιο στην ε, Κομισιόν, διότι πιστεύω ότι εκεί ε, είναι ε, που οι πρωτοβουλίες, ε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να γίνονται και πάντοτε τονίζω ότι πέρα από το έργο που κάνετε εσείς πιστεύω ότι η θέση σας είναι αστεία κατά τρόπο διότι δεν υπάρχει νομοθετική εξουσία αλλά ούτε και δεν φέρετε κάποια ευθύνη θα προκαλέσω λιγάκι λέγοντας ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένη διότι έχει γίνει προβλέψιμο πλέον ότι κάθε φορά που θα συναντώμαστε εδώ πέρα καλείται να για, περισσότερα, ε, για περισσότερες εξουσίες, για περισσότερη συλλογή δεδομένων και το ταυτόχρονα να διαμαρτύρεστε για, τα, ε, για τους περιορισμούς που σας θέτει η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων. Ε, Περιμένω λοιπόν από κάποιον ο οποίος μιλά για την, για την αντιδρομοκρατία να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και να σέβεται περισσότερο τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια αγνοείται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ισορροπία. Ο Επίτροπος Κίνγκ κατά την ακρόασή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή και αυτό είναι το σημαντικό διότι περνάμε τη μία νομοθεσία μετά την άλλη σε αυτό το κοινοβούλιο όμως όταν το ζήτημα αφορά την εφαρμογή τότε βλέπουμε ελάχιστη πρόοδο. Και έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ένα αφορά ε, προς ε, το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο. Έστειλα και γραπτός αλλά και προφορικά ένα ερώτημα Πού βρισκόμαστε λοιπόν ε, στην εφαρμογή της οδηγίας έξι μήνες μετά την ε, εφαρμογή της. Δύο χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν την νομοθεσία και αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πίεση ε, που αισθανθήκαμε όταν έπρεπε να την ψηφίσουμε. Τώρα όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων, ε, βλέπω ότι μοιράζεστε την βελτίωση της ε, ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Όμως προσωπικά ανησυχώ διότι το μόνο για το οποίο φαίνεται ότι συζητάμε είναι το ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας στην Κομισιόν στην οποία συμμετέχετε, υπάρχουν ομάδες και βλέπουμε κάποιες ενδιαφέρουσες αλλά ανησυχητικές πρωτοβουλίες όπου ε, αναφέρεται να δημιουργήσουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων που το αποκαλέσατε εσείς ως ε, το ενιαίο αποθηκευτήριο δεδομένων Και στο έγγραφο δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε θέματα όπως ε, ο δημοκρατικός έλεγχος, ο δικαστικός έλεγχος και ούτω καθεξής. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι μιλάτε για τη δημιουργία μιας μεγάλης βάσης δεδομένων χωρίς όμως να υπάρχει κανένας έλεγχος. Θα ήθελα λοιπόν το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ Γιάννα Άλπρετ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κόφε για την ομιλία του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτά που είπε η Σοφή όσον αφορά την εφαρμογή. Σας έβαλαν στη θέση σας ε, τα κράτη-μέλη, όμως το ερώτημα είναι ποιον ακριβώς συντονίζεται, διότι τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν καλούν ώστε να υπάρξει περισσότερο συντονισμός. Εδώ και καιρό. Δηλαδή όχι μόνο περισσότερο συντονισμός, αλλά και να λάβετε κάποια απτά μέτρα και κάποιος θα πρέπει να συντονίζεται εν τέλει. Έχω το, την αίσθηση ότι όλοι θέλουν περισσότερο συντονισμό χωρίς όμως να συντονίζονται και όλοι θέλουν περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, συνομφωνούμε σε αυτό, όμως κανένας δεν θέλει να κάνει αυτή την ανταλλαγή. Έτσι λοιπόν από την πλευρά των κρατών μελών κάποια πράγματα θα πρέπει πραγματικά να αλλάξουν και ε, καθώς προχωρούμε και υιοθετούμε νέα μέτρα ε, θα ήθελα να δω τι γίνεται με την εφαρμογή των όσων έχουν αποφασιστεί. Εδώ στη Λίμπη αλλά και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2014 ε, η οδηγία ε, ευρωπαϊκών ερευνών και τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια για να το εφαρμόσουν. Απέμεινε μισός χρόνος λοιπόν που ε, θέλω να μάθω πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή. Μερικές φορές μιλάω με κράτη-μέλη, με εκπροσώπους κυβερνήσεων και μερικοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτή η οδηγία. Το θέμα λοιπόν εδώ αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, μέτρα, κοινή αναγνώριση ε, μέτρων έρευνας και καλύτερη συνεργασία όσον αφορά την αστυνόμευση και τα δικαστικά ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να δω κάποιο πρόγραμμα πάνω σε αυτό. Κάτι καλό επίσης είναι ότι αναγνωρίζετε τους αριθμούς της Europol σχετικά με τους ε, ύποπτους τρομοκρατίας οι οποίοι σχετίζονται με προηγούμενα εγκλήματα και οι οποίοι είναι γνωστοί στις διοκτικές αρχές. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπω παντού είναι ότι χρειαζόμαστε μέτρα για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών ε, από ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με κανένα έγκλημα και δεν υπάρχει καν υποψία για αυτό και δεν υπάρχει καν ο κίνδυνος ψηφίσαμε τώρα πάνω στην ε, ε, οδηγία ε, European Area. Τα δεδομένα αυτής όμως, ε, αυτής όμως δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα εγκλήματα. Δημιουργούμε νέα μέτρα τα οποία τα ζητούν με τα κράτη-μέλη τα οποία όμως θα πρέπει να αφορούν ανθρώπους που είναι εγκληματίες και όχι ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν και περνούν τα σύνορα. Θα χρειαστούμε μήπως άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ ή και κάτι τέτοιο. Επενδύουμε λοιπόν δισεκατομμύρια διότι η κατι τετοιο επενδυουμε λοιπον δισεκατομμυρια διοτι η οποία ανέφερε τα συγκεκριμένα δεδομένα καλεί να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα σε ομάδες ερευνών διότι αυτό συμβαίνει κατά τόπους ομάδες οι οποίες, ε, οι οποίες αναζητούν εγκληματίες και πιθανούς ε, τρομοκράτες ε, και οι ντόπιε αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή διότι δεν μπορούν να επενδύσουν άλλο χρήμα ή προσωπικό. Δεν θα ήταν λοιπόν σοφό να θέσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες μας και να μην επενδύουμε σε αυτά τα νέα συστήματα συνεχώς αλλά ανταυτού να πάρουμε χρήματα και να τα επενδύσουμε καλύτερα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της αποκρυπτογράφησης διότι ο υποψήφιος ε, για την ε, θέση στην Κομισιόν ε, για την ασφέλεια είπε ότι υπάρχουν πίσω πόρτες, θα πρέπει να υπάρχουν πίσω πόρτες σε συσκευές αποκριτογράφησης και θεωρώ ότι είναι καλό αυτό. Όμως ταυτόχρονα χάνουμε το στόχο μας διότι αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις καθημερινές μας ζωές. Δεν υπήρξε ποτέ εποχή στην ιστορία που δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για όλους μας. Δεν θα ήταν καλύτερο λοιπόν... Δεν είναι μήπως το πρόβλημα ότι δεν έχουμε το προσωπικό αλλά και τους εκπαιδευμένους ανθρώπους για να μπουν σε αυτά τα δεδομένα ή να κάνουν έρευνες ούτως ώστε να μπουν στα δίκτυα, να ακολουθήσουν τις επαφές και ούτω καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθούμε και εδώ διαφορετικά. Σας Ευχαριστώ. Ο Πίτερ Νίδερμιλερ. Ευχαριστώ κύριε Κύρχοβ για την παρουσίασή σας. Πολύ σύντομα. Αναφερθήκατε αρκετές φορές στη σημασία της προστασίας των σύνορων, τους ελέγχους των σύνορων. Όσον αφορά την ασφάλεια, είναι καθοριστικό το σημείο αυτό του ελέγχου στα σύνορα. Το θέμα όμως της πρόληψης σε μία φράση είπατε κάτι πολύ σημαντικό, μαζική επένδυση και προσπάθεια στην πρόληψη. Αυτό είναι κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μπορείτε να μας πείτε όμως στην πράξη πώς αυτό μπορεί να συμβεί. Πρόεδρος, πρέπει να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο των ερωτήσεων. Να είστε στον κατάλογο εσείς. Γκόμες, Ράζε, Κράντετ. Μπόνι, Βάγκμεντ, Κιάνγκε και Βάινμπεκ. Και κλείνει ο κατάλογος. Άννα μα. Κύριε Δικέρκοφ, καλώς ορίσατε. Μιλήσατε για την αλλαγή του τρόπου δραστηριοποίησης του Μόντου Σομπεράντι και μιλήσατε και για τα χημικά όπλα, αλλά και τα εκρηκτικά σε αυτοκίνητα. Μπορείτε να μας πείτε, παραδείγματο χάρη, πώς είναι δυνατόν να αποφύγουμε κάτι τέτοιο που σήμερα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό να δημιουργήσει κανείς μια τέτοια έκρηξη, παραδείγματο χάρη σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να αγοραστούν αυτά στο ίντερνετ και πάρα πολύ απλά ακόμα και σε σούπερ μάρκετ. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται τέτοιος εξοπλισμός όπως και η μόμπρος διασποράς. Είναι κάτι το εξαιρετικά ανησυχητικό και δεν θα αναφερθώ σε άλλου είδους ανησυχητικά γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν, όπως επιθέσεις κατά πυρηνικών μονάδων. Μιλάτε για ασφάλεια. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατεύσει κανείς τα σύνορα, αλλά πώς είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να μιλάμε για ασφάλεια στα σύνορα, ενώ Κανείς δεν ανησυχεί για τους ασυνόδευτους ανήλικους, τα παιδιά τα οποία έχουν εξαφανιστεί στο εσωτερικό της Ευρώπης, ενώ πρόκειται για άτομα που ήδη έχουν μπει στην Ευρώπη, βρίσκονται στην Ευρώπη, σε καταβλισμούς στην Ελλάδα, αλλού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα άτομα είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Εμείς δεν ξέρουμε πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί, που βρίσκονται. Αφήνουμε τα δίχτυα των διακινητών ανενόχλητα. Και το θέμα του PNR. Το PNR. Ε, ακούσατε την ερώτηση της ε, Σοφή για το PNR. Αλλά εξηγήστε μου τι ακριβώς έλεγχος γίνεται για κάθε είδους ε, λίστες, ε, ονομαστικές λίστες επιβατών και ιδιαίτερα για τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να μεταφερθούν τόνοι από εκρηκτικά, από όπλα, καθότι δεν υπάρχει κανένας είδους έλεγχος, κανένα PNR που να ισχύει για τις ιδιωτικές πτήσεις. Μιλήσατε επίσης για αυτές τις μαζικές επενδύσεις στην πρόληψη. Υπάρχει σήμερα, παραδείγματος χάρη, ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση των ημάμ, των ημάμιδων στην Ευρώπη. Και υπάρχει κάποια δυνατότητα να ενσωματώσουμε την μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρώπη σε όλη αυτή την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσατε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την προπαγάνδα, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών. Μπορείτε να μας πείτε η συνεργασία με τις εταιρείες και τους φορείς παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ έχει προχωρήσει, σε ποιο σημείο βρίσκεται για την καταπολέμηση του, της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ κύριο Στράντε. Σας ευχαριστώ. Τους τελευταίους μήνες διαπιστώνουμε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις τύχησαν ε, πολλές ε, ζωές αθών Ευρωπαίων ε, πολιτών. Βλέπουμε ότι προετοιμάζονται όμως και νέστε τις επιθέσεις από πολύ νέους μαχητές, 15 ετών πολλές φορές. Οι γερμανικές αρχές πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι πολλοί φοβούνται ότι μεταξύ των μεταναστών υπάρχουν και των προσφύγων υπάρχουν σήμερα τέτοιοι επίδοξοι τρομοκράτες. Στην Βουλγαρία όλοι αυτοί οι οποίοι περνάνε ανενόχλητοι από τα εξωτερικά σύνορα μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι δεν ε, περνάνε μαζί τους και τρομοκράτες. Ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι μεταξύ των μεταναστών παρεμποδίζονται οι τρομοκράτες. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο ψήφισμα των ε, Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την κατάρτιση και την καθοδήγηση για να προβλέψουμε μελλοντικές τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι κάνουμε ακριβώς στα αεροδρόμια, τι μέτρα πρέπει να υιοθετηθούν έτσι ώστε να προλάβουμε τέτοιου είδους επιθέσεις στα αεροδρόμια. Χρειαζόμαστε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεκέρκοφ. Στην παρουσίασή σας μας μιλήσατε για τις επιθέσεις στις μεγάλες πόλεις. Όμως, κάποιοι δήμαρχοι μικρών πόλεων και κομοπόλεων στην χώρα μου, στο Βέλγιο, την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν μία ανακοίνωση που αναφέρονται ακριβώς στις πιθανές επιθέσεις σε μικρές πόλεις, κομοπόλεις, Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης τους, που τα μέσα λείπουν. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Αν έχετε συμβουλές, αν έχετε συστάσεις, μιλήσατε για διαφορετικά modus operandi. Ξέρετε σήμερα πώς ακριβώς μπορούμε να προστατευτούμε, υπάρχει ο κίνδυνος επιθέσεων με χημικά όπλα, τι προτείνετε για αυτούς τους μικρούς δήμους, τις κοινότητες, οι οποίοι σήμερα νιώθουν πολύ ευάλωτοι. Η ε, κυρία Κέγκη, ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Η πρώτη αφορά τους, τα, τους ασενόδευτους ανήλικους. Υπάρχει κάποια στρατηγική για την προστασία αυτών των ασυνόδευτων ανηλίκων που πέφτουν θύματα των ε, δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και πολλοί εξαφανίζονται με την άφηξή τους στην Ευρωπαϊκή Επικρότητα. Δηλαδή από ευάλωτη και αδύναμη ε, πρόσφυγες ε, πολλές φορές αποτελούν και γόνιμο έδαφος για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, τα παιδιά αυτά ως εμπόρευμα. Υπάρχει συντονισμός και με αυτά όσα γίνονται για την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων και με ποιο τρόπο γίνεται ο συντονισμό. Και το θέμα τη ένταξη. Υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο. Γιατί γνωρίζουμε ότι εκεί που οι άνθρωποι εγκαταλείπονται στη μοίρα του και στη μοναξιά του, μπορεί πολλέ φορέ αυτό να οδηγήσει και σε βία. Υπάρχει πολιτική βούληση, αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα, υπάρχει αντίληψη και συνειδητοποίηση αυτού του προβλήματος. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Γουίνμπεργκ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κέρχοπα και Δεν άκουσα την αρχική σας εισήγηση. Δυστυχώ καθυστέρησε η πτήση μου. Ωστόσο θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας μέχρι στιγμής και ελπίζω πως όσο γίνεται πιο σύντομα θα μπορέσουν όλα αυτά να εφαρμοστούν κιόλα γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχο του PNR, να ξέρουμε δηλαδή ποιο μπαίνει και ποιο βγαίνει στι χώρε μα. Ε, με την Αναγκόμες επισκεφθήκαμε στην ε, διάφορες χώρες την περασμένη εβδομάδα και είδαμε στα εξωτερικά σύνορα ε, πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να ελέγχονται στο Μάλμε. Έχουμε τώρα μία πόλη που καίγεται. 35 αυτοκίνητα κάηκαν πρόσφατα και μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθεί και χειροβομβίδες. Ε, Ε, διάβασα κύριε Κέργοβ ότι είναι μάλλον απίθανο να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη μετανάστευση και την τρομοκρατία σε κάποια παλιότερη σας συνέντευξη. Εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους τρομοκράτες και τους ε, μετανάστες γιατί βλέπουμε κόσμο που έρχεται με τα βάρκες και μετά κάνει ε, τρομοκρατικές ενέργειες στην Τινησία ή στο Βέλγιο. Είναι πραγματικά ανησυχητικό αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ένα ολόκληρο κατάλογο με τρομοκρατικές επιθέσεις και αυτό συνέχεια μακραίνει. Γι' αυτό και θα ήθελα τα πράγματα να είναι σε γάθαρα. Πρέπει να ενεργήσουμε δραστικά για να σταματήσουν οι τρομοκρατικές ενέργειες. Ευχαριστώ συνάδελφοι πολλές ερωτήσεις. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον μας για αυτό το θέμα. Βασικά, ε, πώς γίνεται ο συντονισμός ανάμεσα στα ε, κράτη-μέλη, γιατί βεβαίως υπάρχει ε, βιασύνη για την εφαρμογή όλων αυτών των δράσεων και για συντονισμό. Πολλές ερωτήσεις. Αν μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα θέματα για να μας απαντήσετε γιατί τέθησαν πολλά σοβαρά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω με αυτό που μόλις είπατε. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ε, εργασία σας κύριε που σε αυτή την Επιτροπή. Είχα τη χαρά ε, να παρακολουθήσω ένα σωρό ακροάσεις και να προσπαθήσω κάθε φορά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Επίσης ήταν εξαιρετικό, εξαιρετική εργασία σας μέχρι τώρα. Η δική μου θέση ορίζεται από τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων, όχι από μένα τον ίδιο. Ίσως να είναι παράξενο, αλλά όταν ε, δημιουργήθηκε η θέση αυτή, ε, και μίλησε για τη δυσκολία αυτού τη αυτής της θέσης γιατί δεν πρόκειται για κάποιο θεσμό, δεν έχει καμία εξουσία και ο μόνος τρόπος να επηρεάσει κανείς τα πράγματα είναι να είναι αξιόπιστος, να ε, βασιστεί και να δημιουργήσει την εμπιστοσύνη, να, μάλλον, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών και της Ένωσης και να είναι και δύο βήματα μπροστά. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω ότι έχω πετύχει τα τελευταία 9 ε, χρόνια έχω την επιστήριξη των κρατών μελών τα, στη διάρκεια αυτών των εννέα ετών, αλλά πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη φάση της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που είχαν υπόψη του στα κράτη-μέλη, ή μάλλον οι επικεφαλής των κρατών μελών, είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια αντιτρομοκρατικη δραση δράση βήμα-βήμα. δεν είναι εύκολο, πρέπει αυτό να το ε, κατανοήσετε. Δεν είναι εύκολο να συνδυάσει κανείς διάφορες κοινότητες, ε, ε πληροφορίες, ε, κατασκοπία, διπλωμάτες, Υπουργεία Οικονομικών, ε, αντιτρομοκρατικές και όλα αυτά να τα συνδυάσω. Μεγάλη πρόκληση γιατί και ο τομέας αυτός είναι πολύ νέος για την Ευρώπη. Συχνά αναφέρομαι στο FBI. Το FBI πέρασε 30 ε, χρόνια ο Έντγαρ Χούβερ 30 χρόνια μπόρεσε να επιβα... Ε, σε 30 χρόνια μπόρεσε να επιβάλλει το FBI στην ε, ομοσπονδιακή στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Εμείς δεν είμαστε καν ομοσπονδία και δεν έχουμε αυτή τη δομή και οργάνωση. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένο με το όσο επιτύχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Εάν με ρωτούσατε πού θα ήμασταν σήμερα πριν από πέντε χρόνια, δεν θα είχα επενδύσει ούτε ένα ευρώ. Ε, δεν θα είχα στοιχηματίσει ε, για το τι έχει επιτευχθεί από την άποψη νομοθεσία. Ωστόσο, είναι πολύ, πολύ ευαίσθητο ο τομέα και είμαι βέβαιο όμω ότι του επόμενου μήνε, λόγω του ηγετικού ρόλου που παίζει η Κομισιόν, λόγω των δεξιοτήτων του Τζούλιαν Κίνγκ, και λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί ότι είναι πρώτη ανησυχία των ε, συμπολιτών μας. 82% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια, ακόμα και αν ε, πρέπει να είμαστε ε, συμπληρωματικοί στην ουσία και, ο πρόεδρος Τούσκο και ο πρόεδρος Γιούνκερ το έπιασαν αυτό το νόημα και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε γρήγορα να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Και φυσικά, κυρία Ινετφέλτ, είναι δύσκολο να κρατηθεί η ισορροπία. Δεν έχω τον χρόνο να σχολιάσω τη δήλωσή σας ότι είμαι αντιδημοκράτης και ότι δεν σέβαμε καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είστε υπερβολικοί ε, εγώ ένα χρόνο τη ζωή μου πέρασα συντάσσοντα το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχω περάσει και πολύ χρόνο σε τρίτε χώρε προσπαθώντα να προωθήσω το κράτο δικαίου και το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί θεωρώ πω είναι πολύ σοβαρά συστατικά για την ε, διαδικασία κατά τη ρισοσπαστικοποίηση. Ε, πολύ περισσότερα πετυχαίνουμε προλαμβάνοντα μέσω τη παιδεία και μέσω τη ένταξη, που ήταν και μια από τι ερωτήσει που ακούσαμε. Εάν δεν κάνουμε περισσότερα, θα μπούμε σε πάρα πολύ πολύ αρνητική, ε, αρνητικό ε, ε, κλιμάκωση της ριζοσπαστικοποίησης. Και ο Επίτροπο Αβραμόπουλο ήταν πολύ αφοσιωμένο σε όλα αυτά τα θέματα και είναι όμω σημαντικό που τώρα έχουμε επίτροπο, ειδικά για την ασφάλεια και όπως είπα, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνδυάσουμε όχι μόνο το Digi Home και την Digi Justice, αλλά και τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνο για την απασχόληση, για την παιδεία, για τον πολιτισμό. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν και έχουμε συμφωνούμε ότι και φυσικά είναι προφανές ότι συνεργαζόμαστε εξαιρετικά καλά μαζί και όπως είπα και στον Τζούλια Κίνγκ ελπίζω να μην με χρειάζεται πια η Κομισιόν να έχει ήδη οικοδομήσει την εμπειρογνωμοσύνη της η Κομισιόν να μην χρειάζεται συντονιστής για την αντιτρομοκρατική δράση πια. Τώρα, πολλά ερωτήματα αφορούσαν την εφαρμογή και θα φροντίσω να σας δώσω μια συγκεκριμένη γραπτή απάντηση για την κατάσταση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Αντάλματος Ερεύνης. Δεν ξέρω ε, πόσα κάτι μέλη έχουν περάσει αυτό το μήνυμα, γιατί δεν είμαι απολύτως ενήμερος. Ξέρω ότι υπάρχει στήριξη, ε, δεν ξέρω όμως πώς έχουμε προχωρήσει, θα επανέλθω όμως συντόμως. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μεριάζονται περισσότερες πληροφορίες. Για την ώρα ο ρόλος μου ήταν να προσπαθήσω να τους πείσω και να εντοπίσω το νομικό εμπόδιο, το τεχνικό εμπόδιο και το ψυχολογικό εμπόδιο. Γιατί δεν έδιναν περισσότερα στο ESIS, το Eurodac, το Europol και την Interpol. Και ε, αυτό είχε αντίκτυπο ήδη, αλλά πιθανότατα θα πρέπει να κινηθούμε με τον νόμιμο τρόπο για να επιβάλλουμε περισσότερη ανταλλαγή στοιχείων και αυτό είναι η διαδικασία κατά παράβαση. Για την ώρα όμως έχουμε ήδη σημαντική πρόοδο για την κρυπτογράφηση. Είναι θέμα και ξέρω ότι ο, ο κύριος Άλμπρεχτ έχει εξαφανιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ζήτημα και δεν έχω την απάντηση και έχω και τις ίδιες ανησυχίες. Είμαι υπέρ της ισχυρής όχι μόνο ώστε να εξασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα, γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχει και να υπάρχουν τα δικαιώματα πραγματική ιδιοκτησία κτλ, Αλλά και γι' αυτό ακριβώ και οι Αμερικανοί μέχρι στιγμή δεν έχουν βρει λύση. Αλλά το θέμα υπάρχει και πρέπει να προβληματιστούμε γι' αυτό. Τώρα, ε, μαζικές επενδύσεις στην πρόληψη. Στην εισήγησή μου μίλησα για αποκατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να φτιάξουν προγράμματα. Οι Γάλλοι ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα για αποκατάσταση των όσων έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και που εθελοντικά ε, θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα αποκατάστασης. Είναι όμως το πρώτο. Θέλουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια, αλλά δεν πάει τόσο γρήγορα. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος, πολλές χώρες έχουν αποτελεσματικά προγράμματα ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Έχει γίνει σύνδεση ανάμεσα στις φυλακές και την τρομοκρατία. Και αυτό είναι θέμα από ριζοσπαστικοποίηση και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Ένταξη, παιδεία, ναι, ε, πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη φαντασία. Το έχουμε ήδη αναφέρει. Να ενώσουμε, να συνδέσουμε ένα εκατομμύριο νέους Ευρωπαίους και ένα εκατομμύριο Άραβες ε, μέσω υπολογιστών. Έχει ένα κάποιο κόστος, αλλά γίνεται. Μετά, εκπαίδευση των ημάμιδων. να αναπτύξουμε δηλαδή ένα ευρωπαϊκό Ισλάμ. Και αυτό με τη δημιουργία εδρών Ισλαμικών σπουδών σε πολλά πανεπιστήμια. Συμφωνώ, αλλά και αυτό έχει κόστος και πρέπει να το ε, συζητήσουμε. Για το ίντερνετ. Μέχρι στιγμής ε, από την πλευρά Europol τα δεδομένα είναι τρομερά. Ε, έχουμε 92% ποσοστό εντοπισμού. Θα ήθελα να προχωρήσουμε όμως ένα βήμα περαιτέρω και ε, να παραπέμπουμε παράνομο περιεχόμενο στις εταιρείε, ούτως ώστε αυτές να κάνουν τη δουλειά μόνες τους. Για την ώρα λοιπόν προσπαθούν να εντοπίσουν έναν αλγόριθμο. Δεν υπάρχει ένα σύστημα με τον οποίο η Google μπορεί να αποστείλει μηνύματα ούτως ώστε ε, να εξετάζουν τις παράνομες ιστοσελίδες Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να πούμε από τη ε, χειρονακτική αναφορά στο να γίνεται αυτόματα και στη συνέχεια να αφαιρείται το παράνομο περιεχόμενο. Όσον αφορά τη μετανάστευση, δεν υπονοώ ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε τις ε, ροές προσφύγων ε, ροές προσφύγαν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί Ε, χρησιμοποιείται από ε, αγωνιστές ε, του ΝΤΑΕΣ. Το είδαμε αυτό από τις επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και είδαμε και πρόσφατα τη σύλληψη ανθρώπων στη Γερμανία που χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο. Δεν έχω όμως όλες τις πληροφορίες πάνω σε αυτό. Έχουν χρησιμοποιήσει λοιπόν τα ίδια σημεία εισόδου, ίσως κρυμμένοι στις προσφυγικές ροές. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για τις μικρές πόλεις Όσον αφορά την ε, παρέμβαση, το γνωρίζετε ότι έχουμε το πρόγραμμα Atlas, το οποίο προσπαθεί να συνδέσει τις ε, μονάδες επέμβασης. Ε, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε αυτό και ενθαρρύνω την Κομισιό να το χρηματοδοτήσει περαιτέρω. Έχουμε το νομικό πλαίσιο για να το εφαρμόσουμε αυτό. Αυτή είναι μία απάντηση και δεύτερον πώς μπορούν οι μικρές πόλεις να αναπτύξουν μια πολιτική αποτροπής. Ε, νομίζω ότι ε, σε αυτό το σημείο μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Πολλά γίνονται σε επίπεδο πόλεων ε, στην, στην εξέφραση της καλύτερης ανταπόκρισης. Η Κομισιόν σύντομα θα σας ενημερώσω, θα έχει με ένα ενωμένο σχέδιο δράσεως σχετικά με το CBR το οποίο θα βασίζεται στα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμή στη Συρία και στο Ιράκ. Γνωρίζουμε ότι το ΤΑΕΣ χρησιμοποιεί ε, χημικά όπλα. Ας το εξετάσουμε λοιπόν όλο αυτό δεν είπα ότι θα συμβεί, αλλά λέω ότι υπάρχουν πληροφορίες ε, και τουλάχιστον θα πρέπει να τις λάβουμε πολύ σίγουρα υπόψη μας ε, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πανεδεχόμενο. Όσον αφορά τα κριτήρια για τη βάση δεδομένων, ε, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Ίσως να θυμάστε ότι υπό την Ολλανδική Προεδρία ε, υιοθετήθηκε ένας οδηγός χάρτης ε, σχετικά με το θέμα αυτό τα κράτη-μέλη προσπαθούν να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά κριτήρια σχετικά με το πώς ε, να παράσχουν τα δεδομένα αυτά προς τη Europol και ναι θα σας έλεγα ότι ε, μπορώ να μοιραστώ τα, τα κριτήρια αυτά με όσους ενδιαφέρονται Πιστεύω ότι κάλυψα. Ε, ο πρόεδρος λέει ότι έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα να πω ότι θα δώσετε μια απάντηση σχετικά ε, με το PNR. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να, πούμε, να μπούμε σε αυτό παρά να μπείτε στη διαδικασία να μπείτε στις ερωτήσεις μία-μία. Ε, συνάδελφοι μας τελειώνει ο χρόνος. Αν λοιπόν ε, υπάρχει κάποιο ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμα θα μπορούσατε να μου πείτε όσον αφορά την ΑΣΟ και το PNR. Όλοι ε, θα δώσει γραπτή απάντηση ο κύριος ε, Ντεκέρκοφε. Έθεσα ένα ερώτημα σχετικά με τη βάση δεδομένων. Δεν άκουσα απάντηση. Ίσως να την, ε, να μην την άκουσα, όμως είναι απίστευτο το ότι η οδηγία PNR, η οποία θα ήταν μια οδηγία κλειδί και εσείς δεν μπορείτε να μας πείτε έξι μήνες μετά το, ψήφι, μετά ε, το ψήφισμα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να, να έχουμε μια γραπτή απάντηση πάνω σε αυτό. Και Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια γραπτή απάντηση πάνω σε αυτό. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί, παρακαλώ ε, σημειώστε το μου ε, και θα το μεταβιβάσουμε. Αυτό λοιπόν ε, όλο δείχνει το πόσο τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται πολύ για την εφαρμογή των οδηγιών σε κάθε λοιπόν συνάντηση αναφέρεται, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάν. Ε, ναι, νομοθετούμε, όχι αρκετά, όμως νομοθετούμε και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δούμε να πραγματοποιείται. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και βλέπουμε ε, το ενεργό ενδιαφέρον των κρατών μελών. Ευχαριστούμε λοιπόν για το ΧΑΣ και θα σας παρακαλούσα να ξανάρθετε στο πλαίσιο μιας άλλης ε, συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τα ερωτήματά τους. So um, Συνάδελφοι, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4. Πρόκειται για την ε, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης για την ΆΣΟ. Είπα προηγουμένως, δεν ήσασταν όμως όλοι εδώ, ότι εκτός από την έκθεση αυτή, Γιορτάζουμε σήμερα τα πέντε χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΣΟ. Έχουμε λοιπόν αυτές τις φωτογραφίες, ενώ ο κύριος Νίντερ Μίλλερ παρουσιάζει την έκθεσή του. Μπορείτε να κοιτάξετε αυτές τις εικόνες, υπάρχουν και οι φωτογραφίες στο βάθος της αίθουσας. Όσον αφορά την έκθεση πρόσθηκε για το σχέδιο έκθεσης, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι πρέπει να μακρηγορήσω με την εισαγωγή αυτού του θέματος. Πίτερ, έχει το λόγο για να παρουσιάσει την ε, έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για τη συνεισφορά τους στην εργασία της ε, Επιτροπής για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης, την Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο. Είναι μεγάλη χαραγημένα που μπορώ να παρουσιάσω σήμερα αυτή την έκθεση και βεβαίως κοιτάξτε και τις εικόνες που πραγματικά δείχνουν ε, κάποια στοιχεία από τη δράση της ΕΑΖΟ. Το σύστημα ασύλου των κρατών μελών σήμερα έχει υποστεί τεράστιες πιέσεις και βεβαίως υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από άλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις όπως ακριβώς κάνουν τα κράτη-μέλη. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει στην σύγκληση των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και των προτύπων όσον αφορά το άσυλο, καθώς και την τεχνική υποστήριξη που πρέπει να προσφέρει στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των αρχών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, αλλά και να υλοποιήσουν ε, όλες αυτές τις αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου βρίσκεται στην καρδιά αυτής της προσπάθειας και εδώ χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να ενισχύσει αυτό το σύστημα μέσω του ΕΑΣΟ. Πρέπει σήμερα να ανταποκριθούμε και να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις Βεβαίω με πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό και θα περιοριστώ σε τέσσερις βασικές πτυχές αυτής της έκθεσης. Πρώτον, η ΆΖΟ θα πρέπει να γίνει μια υπηρεσία ευρωπαϊκή που να συνεργάζεται με όλα τα κράτη-μέλη και την ίδια ώρα να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της. Αυτός ήταν ένας από τους κύριους στόχους της έκθεσής μου. Μία υπηρεσία ευρωπαϊκή που να ανταποκρίνεται σε όλα αυτά που απαιτεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου με περισσότερες οικονομικές δυνατότητες και δυνατότητες σε προσωπικό. Θα πρέπει επίσης η ΆΖΟ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, να συνεργαστεί και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσον αφορά τις δραστηριότητές της, αλλά και όσον αφορά το διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες και τη συνεργασία με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, καθότι πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία δεν μπορεί παρά να είναι υποφελής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κρατημέλη, αλλά και για την ΑΖΟ. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει εδώ να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο αφότι συνεργάζονται ήδη με πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητε της υπηρεσίας. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα επιτρέπει σε αυτούς που αιτούν άσυλο να διεκπαιρεώσουν τις δραστηριότητες αυτές ε, βάσει των συστημάτων που διέπουν την ε, δραστηριότητα των ε, υπαλλήλων της υπηρεσίας ΕΑΣΟ. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ασύλου στην Ευρώπη με μία αξιολόγηση κάθε πέντε χρόνια, προτείνω στα κράτη-μέλη, να αξιολογούνται μία φορά κάθε πενταετία βάσει όλων των πτυχών και προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι προληπτική, καθότι μπορεί να υπάρξουν αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν εγκαίρω. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης θα μας δίνει την πραγματική εικόνα της λειτουργίας του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Δεύτερον, μία αξιολόγηση σε ετήσια βάση σε κεντρικό επίπεδο, μια ανάλυση δηλαδή που θα γίνεται από την ίδια την υπηρεσία, καθότι αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην υλοποίηση και την εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών αρχών. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις και βάσει αυτής της ετήσιας ανάλυσης θα πρέπει να δημιουργείται μία έγκαιρη προειδοποίηση στους τομείς αυτούς και στα κράτη-μέλη αυτά όπου υπάρχουν αδυναμίες. Η ανάλυση των πληροφοριών θα καθορίζει τα θέματα αυτά, τα στοιχεία αυτά που θα πρέπει να ε, αλλάξουν, να τροποποιηθούν σε κάποια κράτη-μέλη ή σε κάποιους τομείς της δράσης της υπηρεσίας. Αυτό βεβαίω μπορεί να γίνεται είτε με ίδια πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάποια κράτη-μέλη, αν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη λειτουργία κάποιας πτυχής του συστήματος ασύλου, θα πρέπει να αποφύγουμε να κινδυνεύσει να εμποδιστεί η ορθή λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος. Αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις και τις συστάσεις μου, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί με μεγάλη χαρά θα ακούσω τα δικά σας σχόλια και θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, Πίτερ. Πολύ ολοκληρωμένη η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την ΕΑΖΟ για τα πέντε χρόνια λειτουργίας της. Πρόκειται για μια υπηρεσία που πραγματικά έχει όχι μόνο υλοποιήσει την αποστολή της, αλλά πραγματικά είναι σαφές σήμερα ότι ο ρόλος και η αποστολή της είναι καθοριστικός. Χρειάζεται περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερα μέσα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές και θεσμικά όργανα σίγουρα θα αποφασίσουν να τις δώσουν περισσότερα μέσα, να βελτιώσουν τη δράση της, έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική, πραγματικά ευρωπαϊκή υπηρεσία για το ευρωπαϊκό άσυλο. Αυτών λεχθέντων θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, συνάδελφο, τον Πίτερ Νίτερ Μιλλερ, για το σχέδιο έκθεση που μας παρουσιάζει σήμερα. Πιστεύω ότι οι συναντήσεις που είχαμε μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ επικοδομητικές και εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια που ακούσαμε, καταρχήν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια υπηρεσία που να μπορεί να καθοδηγήσει και να διευθύνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την ίδια ώρα βεβαίως να σέβεται τις εθνικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι καθοριστικό, διότι δεν μπορεί και δεν πρέπει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου να αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες και ότι μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και αυτό το γραφείο θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Χρειάζεται ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών και βεβαίως τον καθοριστικό και καθοδηγητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, την άμεση δράση όταν αυτό απαιτείται καθότι πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται με την απαραίτητη ταχύτητα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει και παρακολούθηση μετά την δράση. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει σύγκληση όσον αφορά τις αποφάσεις για θέματα ασύλου και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μέσω καλών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τους πιο ηγητές, με τον εισηγητή και είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βίκστρομ. Σε ευχαριστώ πολύ Σεσίλια για την παρουσίασή σου την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά πήραμε το λόγο σε ευρωπαϊκή θεσμή. Ήταν μεγάλη μου τιμή που μας εκπροσώπησε σε αυτή την ε, ευκαιρία και πολλά μπορεί να πει κανείς για το τι έγινε. Θα σας ενημερώσω ποιον θέλει αν έχει ερωτήσει. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πίτερ. Αγαπητέ Πίτερ, ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά σου για αυτό το θέμα. Επίση, ε, θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να συγχαρώ θερμά την σχολιάζω για τα πέντε έτη ε, ε, λειτουργία τη και πραγματικά εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον. Όπως ανέφερε ήδη ο Κάρλος Κουέλιο, η Άζο είναι πολύ βασικό και ε, αρχή για μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Τη χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ και ίσως και στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι ο εισηγητής έχει ακολουθήσει σωστό δρόμο στην σύνταξη της έκθεσης του. Είμαστε ε, σύμφωνοι ότι η ΆΖΟ ε, θα πρέπει να είναι μια ένας ισχυρός οργανισμός ασύλου με διευρυμένη και ενισχυμένη εντολή. Επίσης, συμφωνώ με τον Πίτερ ότι θα πρέπει να υπάρχουν στενοί δεσμοί τόσο με τη ΜΚΟ όσο και με την UNHCR, την υπατερμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε. αλλά πρέπει εδώ να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός είναι και θα παραμείνει πραγματικά ανεξάρτητο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Θεωρώ επίσης πως είναι εξίσου σημαντικό τα βασικά στοιχεία όπως η παρακολούθηση των συστημάτων των κρατών μελών θα διασφαλιστούν και θα ενισχυθούν. Ο εισηγητής για τον κανονισμό του Δουβλίνου θα πρέπει να πω ότι είναι υπεύθυνο αυτός ο οργανισμός για πολλά πράγματα και σε σχέση με το νέο σύστημα επανεγκατάστασης κατάσταση, αλλά θα πρέπει αυτό να το αναλύσουμε πολύ προσεκτικά, καθώς και τις υπόλοιπες προτάσεις που είναι επιτάπητος, όπως η οδηγία περί διαδικασίας, η οδηγία περί δεξιοτήτων, η οδηγία περί ε, συνθήκων υποδοχής που συνδέονται μεταξύ τους. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε με την κάθε μια χωριστά. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την προσέγγιση όπου το Κοινοβούλιο θα εξετάζει όλες τις εκθέσεις για τη μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου σε ένα πακέτο πάνω κάτω, πράγμα που βεβαίως υπερλαμβάνει και την πρόταση ΕΑΖΟ. Το σύστημα θα οριστεί ε, μια φορά όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η εργασία και για να το πετύχουμε αυτό όλοι μας που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το ντοσιέ θα πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τις ε, διάφορες ε, συνάφειες και ε, δεσμούς. Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν εις βάθος συζητήσει με τους συναδέλφους σε διάφορες συνδυασμούς θα ήθελα να ζητήσω σε, αυτή την ευκαιρία μια πρόταση για παράταση της ε, προθέσμιας υποβολής τροπολογιών, αν γίνεται μέχρι τα μέση Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες δηλαδή ακόμα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε και να συντονίσουμε ανάμεσα στους διάφορους εισηγητές ε, τα πράγματα για αυτή τη μεταρρύθμιση. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις επιτάπητος. Ε, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό έργο είναι να μελετήσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες προς αυτή την πολύ καλή έκθεση, που είναι ήδη πολύ καλή. Και επειδή δεν έχουμε άλλα σχέδια εκθέσεων, δεν νομίζω πως μια τέτοια παράταση θα προκαλέσει πρόβλημα για οποιονδήποτε. Προχωρούμε μαζί όλοι. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Ζητώ λοιπόν από τη Γραμματεία να το σημειώσει αυτό προσεκτικά για να εξασφαλίσει πως θα έχουμε χρόνο να σκεφτούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες στις διάφορες ομάδες καθώς και την ε, συσχέτιση ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις. Ευχαριστώ και πάλι, Πίτερ, για την εξαιρετική σου δουλειά και προς την ΕΑΖΟ συγχαρητήρια. 11 Οκτωβρίου είναι για την ώρα η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Να σκεφτεί λοιπόν η στην πρόταση αυτή για παράταση της προθεσμίας. Σκιώδης για το ECR. Ο κύριος Σάλατ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Νίτερ για την, το σχέδιο, Νίτερ για την, ε, το σχέδιο έκθεσης. Ο στόχος είναι να δοθεί τεχνική και επιχειρησιακή αρρωγή προς τα κρατη ε, να αυξηθεί η πρακτική συνεργασία και ανταλλαγή των πληροφοριών ανάμεσα στα κρατη η ε, κατάρτιση προσωπικού καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινού συστήματος ασύλου καθώς και τις ε, δυνατότητες υποδοχής των κρατών μελών. Ναι, Εν γέννη, στηρίζουμε ό,τι προσθέτει αξία στα κρατη για να μπορέσουν να διαχειριστούν την προσφυγική κρίση. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια κρίσιμα σημεία της έκθεσης αυτής. Ο εισηγητής σε πολλές από τις τροπολογίες τονίζει το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την προσέγγιση γιατί η πολιτική και η ιδεολογική ουδετερότητα αυτών των οργανισμών συχνά είναι αμφισβητήσιμη και εν πάση περιπτώσει δεν είναι σίγουρη ή Επίσης είναι σημαντικό για το ECR η αρμοδιότητα για την λήψη αποφάσεων περί ασύλου να ε, παραμένει στα κράτη-μέλη, όπως ορίζει και η πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό δεν στηρίζουμε οποιαδήποτε αναφορά σε κοινή επεξεργασία των αιτήσεων από κράτη-μέλη και τον Οργανισμό Ασύλου. Φυσικά είναι επιθυμητό όλα τα κρατημέλη να χρησιμοποιούν τα ίδια στάνταρ και κριτήρια για να αποφεύγεται ε, η επιλογή ε, η δυνατότητα επιλογή. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Επίση, τα συμφέροντα των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία χορήγηση ασύλου, ενώ ταυτόχρονα αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται όχι μόνο από ανθρώπου ε, που πραγματικά το χρειάζονται, αλλά και από αυτού που δεν το χρειάζονται. Γι' αυτό και οι αποφάσει θα πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ενώ φυσικά θα γίνονται σεβαστοί αυτή σύμβαση τη Γενέβη και η σχετική νομοθεσία. Σα ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω σε συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ να κλείσω τον κατάλογο με άλλον ένα συνάδελφο που ζήτησε το λόγο. Αγιάννα Γκόμες, παρακαλώ να είσαι σύντομη. Και εσύ Σεσίλ, ε, παρακαλώ να είστε σύντομε για να ακούσουμε και τον διευθυντή. Και μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι, εγώ θέλω να, πω, να ευχαριστήσω τον Πίτερ. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Τέρη Κάμπρας, δεν σας είδα. Θα σας δώσω το λόγο. Ναι, στηρίζω τα όσα είπε ο Πίτερ Νίντερμούλερ, αλλά και τα όσα είπε ο Κάρλος Κουέλιο και η Σισίλια Βίξτρομα. Και αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι θα πρέπει να, είναι, να θεωρηθεί ως πακέτο, να εξεταστεί ως πακέτο αυτό, αυτή η νομοθεσία. Ξέρω ότι υπάρχουν σχέδια να μειωθεί ή να υποβιβαστεί η ΕΑΖΟ για να ενισχυθούν άλλοι οργανισμοί όπως αυτοί που ασχολούνται με την ασφάλεια και άρα να μην εστιάσουμε την προσοχή στην πολιτική ασύλου. Αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ευχαριστώ Άννα. Η ε, πράσινη κύριο Στερικάμπρας και ζητώ και πάλι συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σύντομα. Εγώ καλωσορίζω την έκθεση του κυρίου Πίτερ Νίντερ Μίλλερ που υπογραμμίζει τον ε, πήγους ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της ΕΑΖΟ, ειδικά όσον αφορά την επιχειρησιακή και τεχνική αρρωγή σε φάσεις αυξημένων προκλήσεων προς ε, συγκεκριμένα ε, κράτη-μέλη. Αυτή τη νέα πρόταση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα απομακρυνθούμε από τις ε, σπασμωδικές και βραχυπρόθεσμες πολιτικές ε, προς μια ε, προσέγγιση στο άσυλο που θα εστιάζει σε στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη προβαίνουν σε δράσεις, αλλά αυτές δεν αρκούν για να προλάβουν ή να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει να βελτιώσουμε την αρμοδιότητες της ΕΑΖΟ ώστε να υπάρχει ένα σύνολο επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που θα μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη. Συνοψίζοντας, με χαρά βλέπω ότι ο Πίτερ Ντελμιουλέρ συμπεριέλαβε κρίσιμα θέματα που μας απασχολούν πολλού, πολύ στην ομάδα μου των Πρασίνων και μιλώ για τις προτάσεις για το μηχανισμό καταγγελιών, την ενίσχυση του Συμβουλευτικού Φόρουμ και τη δημιουργία ε, του ε, ε, αξιωματικού ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίση, η λογοδοσία της ΕΑΖΟ θα πρέπει, θα πρέπει να μα απασχολήσει. Όταν δίνουμε περισσότερε ευθύνε και αρμοδιότητες σε έναν οργανισμό, θα πρέπει αναλογικά να εξασφαλίζουμε και μεγαλύτερα επίπεδα λογοδοσίας. Σας ευχαριστώ, Πίτερ Νίτερ Μολέρα, και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία τέλος. Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Πίτερ και να θυμίζω ότι φέτος το καλοκαίρι κάναμε μια αποστολή στη Μάλτα. Αυτή η αποστολή ήταν εξαιρετικά σημαντική και τις επόμενες ε, μέρες θα σας δώσουμε και την έκθεση σχετικά με αυτή την αποστολή και θα συνοδεύετε και από προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν ε, τον Πίτερ για τη δουλειά που κάνει. Είδαμε τη σημασία της δουλειάς της ΑΖΟ. Θέλησα να να, μιλήσω και εγώ για να δούμε ότι σε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση όπου ζητάμε, δηλαδή να υπάρχει σφαιρική προσέγγιση, πρέπει να σκεφτούμε την πολιτική ασύλου που η ΑΖΟ θα πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα που αφορούν έναν ε, ετούντα άσυλο. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλ. Ε, Πίτα. Έχεις κάποια τελικά σχόλια. Ε, πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις ε, και εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, βγάλουμε την καλύτερη δυνατή έκθεση και φυσικά περιμένουμε τις τροπολογίες και επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε και με την Γραμματεία για το ζήτημα αυτό αλλά και τις προτάσεις της, για τις προτάσεις της Σεσίλια και ίσως θα μπορέσουμε να βρούμε μια ιδανική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε σε καλά χέρια με εσένα και τους ε, σκιώδεις. Ε, θα ήθελα επίσης ε, να πω όπως επίσης είπες Πίτερ, έχουμε τα πέντε χρόνια της ΕΑΣΟ και όλοι σχεδόν από εμά έχουμε μια κάποια ενασχόληση ε, συμβάλλαμε στο μονοπάτι της ΕΑΣΟ εγώ και πολλοί συναδελφοί μου ασχοληθήκαμε με αυτό θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν ο εκτελεστικός διευθυντής ή ο πρόεδρος θα ήθελα να πούν κάποια πράγματα για να κλείσουν τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ίσως κάποιος από, εσά θα ήθελα να πάρει το λόγο. Αρχικά ο διευθυντής. Ναι, πράγματι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, φυσικά λέει ο πρόεδρος. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά και ε, ευχαριστώ προς τον ε, εισηγητή, αλλά και ε, τους λοιπούς ευρωβουλευτές που βλέπω εδώ, πολλά φιλικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή γιορτάζουμε τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας μας. Από πέρσι το Σεπτέμβρη ε, παρουσιάστηκε το ζήτημα των hot spots, ε, το οποίο ήταν ένα ε, ζήτημα πάνω στο οποίο η Άσο δεν είχε καμία εμπειρία. Και από τότε μέχρι και την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας είδαμε μία αύξηση των δράσεων και μπορέσαμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους μεγάλους αριθμούς κατατόπους. Οι φωτογραφίες αυτές και όπως λέγεται μια φωτογραφία ίσον με χιλιάδες λέξεις θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλή ώρα και δεν θα μπορούσα να περιγράψω την κατάσταση καλύτερα από τις φωτογραφίες που βλέπετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για αυτήν την παρουσίαση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε επίσης ε, τον ε, Πίτα Νίντα για τις ε, προσπάθειές, τους, προσπάθειές του για την κατάθεση μιας έκθεσης σχετικά με τη νέα πρόταση για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό, περισσότερα μέσα και πόρους, χρειάζεται να μεγαλώσουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει μια σωστή απάντηση στην κρίση. Η κρίση δεν ήρθε εδώ για μερικούς μήνες, ήρθε για να μείνει και θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, φτάσουμε σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την προσωπική κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις ε, ε, τροπολογίες που πρότεινε. Ε, μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις με την έκθεση. Είναι σημαντικό να ε, διαχειριστούμε μαζί το θέμα και να ακολουθήσουμε την πορεία αυτή. Χαιρετίζω επίσης ε, τις ε, προτάσεις ε, από την Επιτροπή, η οποία προσπαθεί να υποστηρίξει σε πόρους την υπηρεσία μας και πιστεύω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να βρούμε τις προτάσεις και τις αλλαγές σου ώστε ο ρόλος της νέας υπηρεσίας να γίνει ακόμη πιο ισχυρός πριν φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο για την έγκριση της νέας εντολής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον, τον εισηγητή αλλά και την Επιτροπή Λίμπε για την υποστήριξη της επισκέψης, της κοινέ αποστολές, ε, τους διάφορους τρόπους που βρέθηκαν για να υποστηριχθεί το έργο μας. Ο εισηγητής επικεντρώθηκε στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα ήθελα να αναφέρω ιδιαιτέρως την δημιουργία ενός ε, μηχανισμού ε, διαμαρτυριών το οποίο είναι σημαντικό διότι η ΑΣΟ έχει ως στόχο να βοηθά τα κράτη-μέλη να προσεγγίσουν το ζήτημα με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα λοιπόν είναι άρρητα συνδεδεμένα με το έργο που κάνουμε, με την εκπαίδευση, με το κεκτημένο, με τη βελτίωση ε, του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Εάν βρούμε λοιπόν έναν τρόπο ε, να τα συμπεριλάβουμε καλύτερα, ούτως ώστε να βρούμε ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να τα διασφαλίσουμε είναι κάτι το οποίο εμείς πράγματι χαιρετίζουμε. Παρομοίως ε, χαίρομαι ότι ε, οι υπεπιθύσεις μου που δήλωσα πριν μερικές, ε, μερικούς μήνες στη ΛΥΜΠΕ ούτως ώστε να συμπεριληφθεί και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι κάτι που συμπεριλήφθηκε στη συγκεκριμένη έκθεση δίνουμε πόρους, είμαστε πιο ορατοί στο έργο μας και φέτος και του χρόνου όσον αφορά τις συμβουλευτικές μας αλλά και τη περίληψη της κοινωνίας των πολιτών. Προσφάτως ε, στις Βρυξέλλες αλλά και αλλού ε, δημιουργανώσαμε αρκετά εργαστήρια με την κοινωνία των πολιτών ε, και κάτι ακόμα σχετικά με την αύξηση συνεργασίας με την υπατιαρμοστία του ΟΗΕ. Είναι μία δήλωση της πρακτικής ε, έχουμε ένα γραφείο ε, της ΥΠΑ της Αρμοσίτιας εντός της ΕΑΣΟ. Έχουμε εβδομαδιαίες ε, συναντήσεις, ετήσιες αναφορές. Είναι γεγονό λοιπόν ότι όλο αυτό θα φανεί καλύτερα ε, στην νέα νομοθεσία. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το ημερολόγιο το οποίο προτάθηκε από την ε, ΛΥΜΠΕ είναι σημαντικό όσο πιο νωρί το έχουμε και λαμβάνοντας υπόψη ε, τη στιγμή ε, που έχουμε, το momentum θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν ε, για την υποστήριξη που μας δίνετε. Κοιτάζω τον εισηγητή και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την Κομισιόν ώστε να απαντήσει κάποια ερωτήματα. Λυπάμαι όμως που θα δυσαρεστήσω την Κομισιόν αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Ε, μία σύντομη ίσως απάντηση προς τον εισηγητή ίσως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτό και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση και για την πρόοδο καθώς επίσης και το ρυθμό με τον οποίο ε, σκέφτεται να το προωθήσει. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς τον εισηγητή ε, διότι φαίνεται ότι συμφωνεί με την πρόταση της ε, Κομισιόν σε βασικά ζητήματα όπως είναι για παραδείγμα η ε, λειτουργική και η τεχνική βοήθεια. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία τα οποία θα θέλαμε να εξετάσουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως είναι το ζήτημα ε, της εκπαίδευσης, όπου θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία σχετικά με το πώς θα γίνεται η εκπαίδευση, η συνεργασία με την ύπατη αρμοστία, με ΜΚΟ, και αυτά είναι σημαντικά, όμως ε, θα θέλουμε να αναλύσουμε τις τροπολογίες για να το εξετάσουμε καλύτερα. Όσον αφορά τις δικαστικές αρχές, ε, πώς μπορούν να συμμετάσχουν αυτές ε, στην όλη διαδικασία, η εφαρμογή του εκτελεστικού διευθυντή, εκεί ο εισηγητής πρότεινε ε, να υπάρχει κοινή ακολουθία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και αυτό ε, ξεφεύγει λιγάκι από την πρόταση της ε, Κομισιόν. Ανησυχούμε για το ότι η έκθεση ε, προσπαθεί να ε, ξεφύγει από, τις, από τον αριθμό ε, των θητιών που θα μπορεί να έχει ο κάστοτε διευθυντής Και τέλος ε, όσον αφορά ε, τον μηχανισμό διαμαρτυρίας ε, τον, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριφολικής και Ακτοφυλακής και θα θέλαμε να δούμε πώς αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στην υπηρεσία σύλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Νίνταμπελα, τους Σκιώδης, τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε καθώς επίσης σας ευχαριστώ και για την έκθεση. Όπως προαναφέρθηκε η 11η ε, Οκτωβρίου είναι πολύ σύντομα για την κατάθεση τροπολογιών, οπότε θα εξετάσουμε αν μπορεί να παραταθεί. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε μια αιωνιότητα, χρειαζόμαστε μόλις μερικές εβδομάδες ε, και ε, νομίζω ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μας αυτό δεν είναι δυνατό. Α, μπορεί να γίνει μέσω του εισηγητή αυτό. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 που αφορά τι επιπτώσει των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, με διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου. Η συγκήτρια είναι η Άννα Γκόμες. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα, θα δώσω το λόγο λοιπόν στην Άννα μας για να εξηγήσει. Σας ευχαριστώ. Μία εκμάζουσα οικονομία με βάση τα δεδομένα σημαίνει διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, υπηρεσιών και βελτιωμένη παραγωγικότητα. Και για αυτό το λόγο κάποιοι αποκαλούν ε, την συγκεκριμένη υπόθεση τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Βεβαίω είναι μια προοπτική που ήδη έχει εξεταστεί από τους συναδέλφους στην Επιτροπή Ήτρε, αλλά επίσης και στο ψήφισμα που εγκρίθηκε φέτος που αναγνωρίζει ότι πρέπει να, να αναλύσουμε πώς τα big data, τα, που είναι η βάση για αυτή τη βιομηχανική επανάσταση, μπορούν να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, γιατί εκεί περιλαμβάνουν, αυτό σημαίνει μάλλον πολλές προκλήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θεομελιώδη ε, δικαιώματα. Ορισμένοι θεωρούν πως τα big data αφορούν μόνο τις στατιστικές. Επισχυρίζονται ε, ότι είναι απλά στατιστικές που βασίζονται στις τεράστιες βάσεις δεδομένων. Ε, αυτό ας πούμε είπαν κάποιοι ε, στη Silicon Valley όταν που την επισκεφθήκαμε νωρίτερα φέτος, αλλά βεβαίως και δεν πρόκειται για παραδοσιακές στατιστικές ή για απλές βάσεις δεδομένων δεν αυτό επηρεάζει ας πούμε, το δικαίωμα ιδιοκτησίας κατοχής ε, βιομηχανικών δεδομένων. Ε, γιατί εκεί η βάση είναι ατομικά στοιχεία, ατομικά στοιχεία μεμονωμένα τα οποία χρειάζονται προστασία ακόμα και αν αυτά έχουν ε, καταστεί ανώνυμα. Δεδομένες της σταδιακής εσώρευσης στοιχείων των συστημάτων δεδομένων, των βασίων δεδομένων που συλλέγουν διάφορες, ε, διάφορα στοιχεία από διάφορες πηγές, καθίσταται λένε και πιο ε, ε, προφανές ότι η, τα υποκείμενα των στοιχείων γίνονται να γνωρίσουμε και άρα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ασφαλιστικές δικλείδες και γι' αυτό και ε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για αυτό το θέμα και ξέρω για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ ότι την έκθεση FTC και την έκθεση του Λευκού Οίκου για αυτό το θέμα για τη συσχέτιση των big data μαζί με, το, τα, ε, με το ίντερνετ ε, προκαλούν ανησυχία και την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα σε ένα σεμινάριο που οργανώθηκε από τα γερμανικά ε, γερμανικές βιομηχανίες ως εκπρόσωπος της BMW τόνισε το πρόβλημα, ότι, το πρόβλημα της μοιρασιάς, ε, μάλλον της κοινοποίησης στοιχείων, των δικών του στοιχείων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Προσωπικά στοιχεία είναι αυτά. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα εγγύσεων. Συμβαίνει ήδη αυτό το πράγμα, γίνονται αναλύσεις, αλλά με μεγάλο βαθμό αδιαφάνειας. Και φυσικά επικρατεί έλλειψη ε, νομοθεσία σχετικές. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει το άτομο, το υποκείμενο, πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του και δεν μπορεί και να εμπιστευτεί ε, ποιος τα χρησιμοποιεί. Ας πούμε, έχουμε τις, τα, τα, τις συσκευές, τα διάφορα μικροτσίπ και τα λοιπά. Ε, Έχουμε βέβαια παραγωγή συνεχή στοιχείων, αλλά αυτό δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό από τον κόσμο, από τα άτομα. Εγώ μάλιστα βλέπω ε, ότι γίνεται πολύ καλή χρήση κάποιες φορές, μάλλον πο, πολλούς τρόπους όπου θα μπορούσαν τα big data να χρησιμοποιηθούν πολύ θετικά. Όχι μόνο για τη χάραξη πολιτικών, αλλά και για την ε, πιο διαφανή και πιο υπόλογη ε, υπεύθυνη δίκηση. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τρόποι, μέθοδοι που οδηγούν σε profiling και σε άλλα αρνητικά ε, αποτελέσματα που πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και γι' αυτό και χρειάζεται δική μας έκθεση και φυσικά οι συνάδελφοι είμαι βεβαία ότι θα συμβάλλουν σε σύνταξη αυτής της τόσο σημαντικής έκθεσης Πρέπει να εστιάσουμε κατά τη γνώμη μου στην ε, σημασία της διαφάνειας όσον αφορά την χρήση και την αξία της συλλογής των στοιχείων, να διαχειριστούμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και αναλύονται όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς και να δώσουμε στοιχεία στον κόσμο για το πώς γίνεται αυτή η επεξεργασία ή ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το να συνδεθούμε με τη διαφάνεια θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το άτομο έχει τη δυνατότητα να δώσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή για την ανάλυση των στοιχείων του, είτε είναι για την αγορά, είτε είναι για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών ή οτιδήποτε και έτσι να υπάρχουν και άλλες διατάξεις που να μην επιτρέπουν την κατάχρηση στοιχείων χωρίς τη συγκατάθεση των ε, ανθρώπων ε, που τους αφορούν. Να δούμε επίσης πώς θα απαγορεύσουμε τη χρήση των στοιχείων για profiling και για διακρίσεις στην ουσία Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνονται θα, δεν θα οδηγούμαστε σε παράνομες διακρίσεις λόγω της χρήσης όλων αυτών των big data. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Όλοι φαντάζομαι προετοιμαζόμενοι θα διαβάσατε πώς όλα αυτά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δυτικότητά μας. Ε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το θέμα, πολύ σημαντικό και έχουμε μεγάλη πυρογνωμοσύνη εδώ στην Επιτροπή μας για να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Διαπίστωσα ότι και η Επιτροπή Ήτρε θα συντάξει γνωμοδότηση, αλλά με τις άποψεις ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο θέμα του πώς τα πως οι εταιρείε του ίντερνετ παίρνουν τα στοιχεία μας και πώς τα επεξεργάζονται και πώς επηρεάζει αυτό τον ιδιωτικό μας ε, χώρο. ευχαριστώ και ξεκινάμε τον κύριο Βος. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει σίγουρα να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψηφιοποίηση είναι κάτι που μόνο τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Πιστεύουμε, θεωρούμε ότι όλα θα αλλάξουν. Έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάμε για τα μεγάλα δεδομένα, big data, διαπιστώνουμε ότι σίγουρα μπορεί να υπάρξουν κάποιοι κίνδυνοι, κάποιες απειλές, αλλά σίγουρα και κάποιες ευκαιρίες καθότι οι εφαρμογές που απορρέουν από τα big data μπορεί να είναι τεράστιες. Εδώ δεν αφαιρόμαστε μόνο βέβαια στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά στο θέμα του ανταγωνισμού, στις οικονομικές συνέπειες, θέματα ασφάλειας και Βεβαίως ε, σε ατομικό επίπεδο το θέμα της ε, υγείας. Καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις και οι εφαρμογές εδώ μπορεί να είναι πολύ άριθμες. Υπάρχει ο Γενικό κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Το πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του, αλλά πιστεύω ότι εδώ χρειαζόμαστε και κάτι επιπλέον. Ενδεχομένως δηλαδή μια καλύτερη, ευκολότερη πρόσβαση προς αυτά τα δεδομένα, τα οποία ίσως θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και σε καθημερινό επίπεδο. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα και στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με εφαρμογές όπως καταπολέμηση κάποιων ε, ασθενειών. Και μόνο εάν λειτουργήσουμε με αυτό τον τρόπο και μόνο εάν δηλαδή μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά με ένα συγκεκριμένο τρόπο και για πολύ συγκεκριμένες και δεδομένες χρήσεις, Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να μπορεί κάποιος να το ε, ελέγξει, να το αναγνωρίσει. Βεβαίως λοιπόν, ας μην ε, γελιόμαστε, υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία, τα συνειδητοποιούμε χωρίς ακριβώς να ξέρουμε ποιες είναι όλες τους οι επιπτώσεις, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν και οι επιφυλάξεις και οι περιορισμοί, δηλαδή να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε κάποια δεδομένα, αλλά για συγκεκριμένες χρήσης μόνο. Και αυτό βεβαίως χρειάζεται μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση και βεβαίως αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλη χωρίς την ίδια ώρα να περιορίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται. Uh, Ο κύριος Άλμπρεχτ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία βεβαίως είναι στα πλαίσια των πρωτοβουλειών και άλλων ε, επιτροπών που αφορούν ε, το μεγάλο αυτό θέμα, τα big data. Σίγουρα αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε για κάτι το οποίο ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τι είναι big data? Big data είναι ένα password δεν ξέρουμε ακριβώς κανείς από μας περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως το συζητούμε εδώ και καιρό και το θέμα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, τα λεγόμενα smart data. Και αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ είναι να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, ποιες θα είναι οι εφαρμογές και οι επιπτώσεις. Και πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι είναι ίσως καλύτερο να δούμε ποια χρήση μας ενδιαφέρει, τι θέλουμε να κάνουμε. Η συσσόρευση δεδομένων, η αποθήκευσή τους, πολλές φορές οδηγεί σε πολύ αυστηρές ε, κριτικές και ξέρετε ότι αυτό που σήμερα δεν γνωρίζουμε είναι ποια θα μπορούσε να είναι η χρήση όλων αυτών. Για τι ακριβώς μιλάμε όμως. Μιλάμε για προσωπικά δεδομένα. Γιατί εδώ η προστασία των προσωπικών δεδομένων σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να ισχύσει και πολύ πριν αρχίσει να ισχύει αυτή η έκθεση. Και το θέμα βεβαίως της χρήσης, της υλοποίησης των κανόνων, των προτύπων και το δύσκολο, αν θέλετε, είναι να μεταφέρουμε τις γενικές ιδέες και την νομοθεσία που θα προετοιμάσουμε στην ε, πράξη με όλες τις τεχνικές επιπτώσεις. Τα προσωπικά δεδομένα, λοιπόν, τα οποία πολλές φορές... Ε, δεν είναι χρήσιμα για να προχωρήσει κάποιος, ε, παραδείγματο χάνει σε μια καινοτόμα εφαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να ξέρουμε περί πρόκειται, ποια είναι τα δεδομένα που χρειάζονται και βεβαίως όλοι γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά αυτού που θέλουμε να απελευθερώσουμε και να βοηθήσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, την προστασία των έξυπνων διαδικασιών και δεδομένων και βεβαίως να απλοποιήσουμε και να μειώσουμε τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση. Επίσης θα πρέπει να επανέλθω και εγώ σε αυτό που είπε η Άννα Γκόμες, το θέμα των ε, διακρίσεων. Δηλαδή, οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ακόμα λοιπόν και αν ε, δέχονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την παραχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν καταλαβαίνουν, παραδείγματος χάρη, τι ακριβώς, ε, σε τι ακριβώς ανταποκρίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, οι αλγόριθμοι. Γι' αυτό και κοιτώντας τα σημερινά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πιο απλές, πιο διαφανείς διαδικασίες, ιδιαίτερα για όλες αυτές τις εφαρμογές, τις οποίες ε, καθημερινά καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε περιεχόμενο, παραδείγματος χάρη στο ίντερνετ κτλ. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, Νομίζω θα πρέπει να βάλουμε και κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες δεοντολογίας. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα δεδομένα που μπορούν να ενσωματωθούν στην ανάλυση των big data και ποια όχι. Μπορούμε να τα ενσωματώσουμε όλα. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση όσον αφορά την παράμετρο ασφαλείας των κοκκινομάλιδων. Πρέπει να τα αναλύουμε όλα. Ναι, ίσως θα πρέπει καταρχήν να επιλέξουμε τις αναλύσεις αυτές που θέλουμε να γίνονται και να βάλουμε και κάποια όρια. Να πούμε δηλαδή ότι κάποιοι τομείς μπορεί να αναλύονται, αλλά εντελώς ανώνυμα, παραδείγματο χάρη. Αυτή είναι και η δική μου συνεισφορά και θα ήθελα στο μέλλον να ενσωματωθούν αυτά τα σχόλια. Mrs. Stevens, please. Dankjewel, voorzitter en collega's. Ik zal het kort houden ook. Ik wil graag de verslaggever bedanken voor de Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την παρουσίασή της. Πιστεύω ότι θα πρέπει σίγουρα να μπούμε στο βάθος αυτής της ανάλυσης εξετάζοντας τις απειλές και τα πλεονεκτήματα. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία, να προστατεύσουμε την καινοτομία. Τα big data είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, έχοντας όμως πάντα κατά νου την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ναι, να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα, χωρίς να ξεχνάμε την προστασία της, προσ... της ιδιωτικής ε, ζωής. Ποια είναι τα όρια όσον αφορά την ε, ανάλυση των δεδομένων. Μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά που μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας. Και ποια αποκλείονται. Όλα τα δεδομένα. Ποιος κάνει τον έλεγχο. Ποια είναι η εποπτική αρχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στη συζήτηση δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο των κρατών, των εθνικών κρατών, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ βρισκόμαστε απέναντι στους ε, γίγαντες, στο Twitter, στο Amazon, Google. Ξέρετε ότι το Facebook έγινε ε, αντικείμενο λογοκρισίας πριν από λίγο καιρό και αυτό βεβαίως είναι περιορισμός στην ελευθερία έκφρασης. Πώς λοιπόν μπορούμε εδώ να εγγυηθούμε σε κάθε περίπτωση την ελευθερία έκφρασης. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση όταν μιλάμε για τα big data και την επεξεργασία των δεδομένων. Εγώ θα συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι ιδιαίτερα για την συνεργασία που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λόρισταν. Thank you Ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι που ήδη ακούστηκε. Ο κανονισμός ε, για την ε, προστασία των γενικών δεδομένων είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτησή μας και πιστεύω θα πρέπει από εδώ και πέρα να βρούμε τρόπους να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή. Κοιτάξτε, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ σήμερα δεν είναι απλοί ηλεκτρικοί, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Πρόκειται για κάτι το οποίο κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από την επεξεργασία των δεδομένων. Είναι σαν να συγκρίνουμε τον ψηφιακό κόσμο με τον ε, κόσμο τον αναλογικό. Και οι ανησυχίες του κόσμου προέρχονται από ακριβώς αυτό. Εδώ μιλάμε για την ανάλυση των δεδομένων, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας και της ανάλυσης και η εφαρμογή, η χρήση τους αυτών των αποτελεσμάτων. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι ε, για όλους μας. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν. που αφορούν ακριβώς αυτήν την ανάλυση των big data. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί από την υπάρχουσα νομοθεσία από τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πώς οι δυνάμεις, και σε αυτές συμπεριλαμβάνω και τις οικονομικές δυνάμεις, θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και αυτή την ανάλυση. Και σκοπός μας εδώ εμάς των πολιτικών αρχών είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από αυτές τις δυνάμεις. Έχουμε λοιπόν ήδη αρκετή εμπειρογνωμοσύνη και είναι σημαντικό να κατευθυνθούμε προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν πρέπει εδώ να αρχίσουμε μια τεχνολογική συζήτηση. Αυτό πρέπει να γίνει κάπου αλλού, όχι εδώ. Μια τελική παρατήρηση θα ήθελα να κάνω πριν δώσω το λόγο στην Άννα Γκόμες. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε διαβάσει αυτά τα συμπεράσματα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω για την έκθεση είναι ότι Σίγουρα το πλαίσιο συνεχίζει να είναι ο κανονισμός και ενώ πρόκειται για έκθεση ιδέες πρωτοβουλίας θα πρέπει να παραμείνουμε εντός αυτού του πλαισίου. Ξέρετε ότι οι εξελίξεις ε, είναι ταχύτατες στον τομέα αυτό, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε σε κάποια σημεία συμβουλές εμπειρογνωμόνων. το θέμα της αλληλεπίδρασης αυτών των δεδομένων στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιος όγκος προσωπικών δεδομένων, πολύ προσωπικών δεδομένων του καθενός από εμάς στο διαδίκτυο. Και σαφώς οι περισσότερες ανησυχίες για την έλλειψη προστασίας της ιδιωτικής ζωής ε, σίγουρα προέρχεται από αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδομένων. Σίγουρα λοιπόν εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή μοντέλου θα έλεγα και βεβαίως ε, σε αυτό εμπλέκονται και οι μεγάλοι γίγαντες ε, Google και άλλες επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ακούσουμε και κάποιους εμπειρογνώμονες, να δούμε ποιες είναι οι δικές τους προσεγγίσεις. Σίγουρα όμως αυτή η έκθεση θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά τους. Τον Γιάννα και την ε, Μαρία Λόρισιν που μπήκαν στην ουσία. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή και να μιλήσουμε για την τεχνολογία. Ξέρουμε που βρισκόμαστε και όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε αυτή την προστασία, να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει και αυτό από τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις, παραδείγματο χάρη, που ανταλλάσσουν δεδομένα, ανταλλάσσουν βάσεις δεδομένων, παίρνουν αποφάσεις βάσει των δεδομένων που συλλέγουν και των αναλύσεων αυτών και δεν ε, ενδιαφέρονται καθόλου για το GDPR. Και αυτό βεβαίως ε, ισχύει και για όλους τους φορείς που χειρίζονται big data οι οποίοι βεβαίως δέχονται ότι αυτοί οι κανόνες και το GDPR σίγουρα δημιούργησε κάποια, ένα νέο ε, πλαίσιο, μια ασφάλεια, μια βεβαιότητα, εκεί που εκείνοι δεν ήθελαν κανένα κανόνα. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι τις αφήνουμε προς χρήση. και πολλές φορές ε, ε, δεν το υποψιαζόμαστε καν ότι τόσο προσωπικά δεδομένα, δεδομένα για την υγεία μας, άνθρωποι παραδείγματος χάρη, ε, που πάσχουν από πολύ σοβαρές ασθένειες και βρίσκονται και στο τελικό στάδιο, τα δεδομένα αυτά πολλές φορές μπορεί να μεταφερθούν. Καταλαβαίνετε ότι η ανάλυση αυτών των δεδομένων, ότι η πληροφορίες που παρέχονται ακόμα και από τα δίκτυα ενέργειας, πράγματι, δεν είναι ουδέτερες πληροφορίες, δεν είναι ουδέτερα δεδομένα. Και βεβαίως βλέπουμε σήμερα ότι η χρήση αυτών των δεδομένων μπορεί να γίνεται και από νέα παιδιά που εργάζονται και στην Καλιφόρνια κάνουν κώδικα χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν σήμερα τεράστιες κεφαιρίες και τεράστιες δυνατότητες και σίγουρα θα περιοριστούμε στο πλαίσιο του κανονισμού. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο, που είναι η ανταλλαγή στην υπόφωνη των DNA με τη Δανία. Εδώ θα παρουσιαστούν τα δεδομένα από όλα τα κράτη που συμμετέχουν και βεβαίως η γνωμοδότηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες. Έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε την απλοποιημένη διαδικασία παρουσίαση και κατόπιν σχέδιο έκθεσης. Σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να παρουσιάσετε το θέμα σας πολύ πολύ σύντομα okay, I feel rather foolish uh, having gone through that whole thing without them not being here. It's difficult in this bigger room. Ο εισηγητή δεν είναι εδώ. Είναι δύσκολο να δούμε σε ένα τόσο μεγάλο δωμάτιο, σε μια τόσο μεγάλη αίθουσα, ποιο είναι και ποιο δεν είναι. Έχουμε την ψηφοφορία που του περούν στα σημεία 8 και 9. Μπορούμε να περάσουμε εκεί. Γνωρίζει κανείς που είναι η Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ε, θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για την ε, πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου ε, σχετικά με την ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών στοιχείων και στοιχείων δεδομένων. Τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την ε, γενική διάταξη σχετικά με την προστασία δεδομένων στο κεφάλαιο 6 της απόφασης 2008 635 ΔΕΗ σύμφωνα με το οποίο αυτό αποτελεί ε, προϋπόθεση για την ανταλλαγή ε, δεδομένων και την ανταλλαγή δεδομένων ε, δακτυλοσκοπικών στοιχείων. Η Γραμματεία του Συμβουλίου υπο, κατέθεσε στις 19 Αυγούστου την απόφαση ε, για τη Δανία ώστε να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο κάλεσε το ε, Κοινοβούλιο να παρουσιάσει μέσω ψηφοφορίας εντός τριών μηνών, την απόφαση της. Και όλο αυτό σε σχέση ε, αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διασυνοριακής εγκληματικότητας και παρακαλούμε το Κοινοβούλιο να καταθέσει την απόφαση του όσο δυνατόν γρηγορότερα για την εφαρμογή της συγκεκριμένη απόφασης. Ευχαριστώ πολύ και όπως προανέφερα οι συντονιστές αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό στο πλαίσιο προποιημένης διαδικασίας και θα ψηφίσουν πάνω σε αυτή την έκθεση. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στα σημεία 8 και 9, το οποίο αφορά τη συμφωνία και επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και της Ευρωπόλου, ενώ το 9 τη συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλου. Είναι μια συμφωνία που κινού μεταξύ της Προεδρίας, και του, Συμβουλίου, της Προεδρίας του Συμβουλίου και της ε, θεωρούν ότι οι συμφωνίες που περιλαμβάνουν επίσης ε, και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων και γι' αυτό το λόγο αποτελείται έγκριση. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η συνεργασία της Europol ε, περιλαμβάνεται ακόμα στον τρίτο πυλώνο, πυλώνο όπου καλείται η ε, γνώμη της, του Κοινοβουλίου και μας δίνεται περιορισμένος χρόνος για να αποφασίσουμε αυτό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ακολουθήσουμε επιτυχημένη διαδικασία. Κάποιοι ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό θα εφαρμοστεί από το Μάιο. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου αλλά και στον εκπρόσωπο της Ευρωπόλ για να παρουσιάσει αυτές τις συμφωνίες και τις ε, λειτουργικές ανάγκες για όλο αυτό και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο για ερωτήσεις και σχόλια αρχικά ο κύριος Μπαράν από την Σλοβακική Προεδρία και στη συνέχεια ο κύριος Νιούμαν από την Ευρωπόλ. Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ε, συμφωνίες ε, για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και ε, Ευρωπόλ, αλλά και Γεωργίας Ευρωπόλ. Δεν είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία, θα γνωρίζετε τη διαδικασία. Η Ευρωπόλ κάνει αίτημα προς το Συμβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή μιας τέτοιας συνεργασίας με τρίτη χώρα. Ε, στη συνέχεια λαμβάνοντας την γνώμη του Κοινοβουλίου αλλά και του Υποπτικού Συμβουλίου το Συμβούλιο εγκρίνει επιτρέποντας την Ευρωπόλ να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Όσον αφορά την ίδια τη συμφωνία, η Ουκρανία είναι ένας ε, σημαντικός εταίρος ε, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας αλλά και της ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης υπάρχουν νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις ε, Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται από την Συμφωνία Σύνδεσης το οποίο εγκρίθηκε το 2014 αποτελεί μια νέα, ε, μια νέα κατάσταση στις σχέσεις Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την πολιτική σύνδεση αλλά και την οικονομική ολοκλήρωση. Παρέχει την δέσμευση ε, για εγκύτερες σχέσεις με βάση τις ε, κοινέ σχέσεις και σεβασμό προς ε, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η η Ευρώπη και η Ουκρανία συνεργάζονται τη βάση μιας στρατηγικής ε, συμφωνίας που υπογράφηκε κατά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας το 2009. Στόχος είναι να υπάρχει μια επιχειρησιακή συνεργασία για το 2011 και στη συνέχεια η ε, μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων ξεκίνησε ο βασικός στόχος ε, για την προστασία δεδομένων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Το Εποπτικό Συμβούλιο ε, δίνει την άδεια στο Διευθυντή της Ευρωπόλου να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την, με την Ουκρανία για την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή είναι επίσης σημαντική διότι η συμφωνία είναι μία από τις υποχρεώσεις για την απελευθέρωση των θεωρου... θεωρήσεων των Ουκρανών. Μία συμφωνία μεταξύ της Ευρωπόλ και της ε, Γεωργίας ε, καθοδηγείται από τις κοινέ αξίες, τις κοινές αξίες, τη σταθερότητα στην Γεωργία, αλλά και τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ούτω ώστε να υπάρξουν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία υπέγραψαν μια συμφωνία σύνδεσης η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2016 και έχει ως στόχο να εμβαθύνει τις ε, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχοντας υπογράψει, έχοντας τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γεωργία έχει αναλάβει υποχρεώσεις στους τομείς της ε, δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, ε, θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, η συμφωνία δεσμεύει την γεωργία ούτως ώστε να προβεί σε μεταρρυθμίσεις όπως είναι το εμπόριο, η οικονομική επανόρθωση και την διακυβέρνηση προσφέροντας δυνατότητες συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή καθ' αυτή είναι αποτέλεσμα ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας. Η Γεωργία είναι μία από τις 16 χώρες εταίρους Τον Ιούλιο του 2016 το Εποπτικό Συμβούλιο εξέδωσε μια θετική γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου από την Ευρωπόλ και ο οποίος θα σας παρουσιάσει τους επιχειρησιακούς λόγους για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θα, ήθελα να, θα θέλαμε να εμβαθύνουμε τη επιχειρησιακή μας συνεργασία με την Ουκρανία και τη Γεωργία αφορά διάφορους τομείς εγκλημάτων όπως τα οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα σχετικά με ναρκωτικά, κάποιοι, κάποιοι τομείς που θα ήθελα να τονίσω αφορά τις ε, κινητές ε, οργανωμένες ομάδες εγκλήματος που είναι ενεργές ε, σε οργανωμένες κλοπές, σε ένοπλες κλοπές και ούτω καθεξής. Και μέχρι στιγμής η συνεργασία που είχαμε με τη Γεωργία ήταν όσον αφορά την ανταλλαγή μη προσωπικών δεδομένων και τώρα θα θέλουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίε όχι μόνο για τα εγκλήματα αλλά και του εγκληματίε, Επίσης όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων θα θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ουκρανία καθώς η Ουκρανία ε, είναι χώρα ε, μετάβασης. Ε, μιλάμε για τις χερσαίες οδούς στα σύνορα της Ουκρανίας και σύμφωνα με τα με τις πληροφορίες μας πρόκειται, έχουμε ακόμα και Ουκρανούς διακινητές Τέλος, έχουμε υποφεληθεί από τις ε, πολύ καλές ε, συνεισφορές από την αστυνομία της Ουκρανίας σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα γενικότερα και έχουμε ταυτοποιήσει ε, και άλλους σύνδεσμους μεταξύ κρατομελών και τις έρευνες που κάνουν αλλά και την Ουκρανία και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε να έχουμε ε, πολύ καλές πληροφορίες ε, τώρα όσον αφορά τη γεωργία ε, και εκεί θα θέλαμε να νοικοδομήσουμε, να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας, όπως είναι για παράδειγμα στον τομέα της τρομοκρατίας. Η Γεωργία χρησιμοποιείται ως χώρα μετάβασης για ξένους μαχητές από την περιοχή του Κάφκασου Πολλοί λοιπόν μεταβαίνουν στις περιοχές μέσω της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν και οι αρχές της Γεωργίας είναι διατεθειμένες να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους αγωνιστές. Όσον αφορά την Γεωργία υπάρχουν επίσης πολλοί τομείς όπου θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Ένας τομέα που θα ήθελα να τονίσω αφορά να αγωνιστούμε από κοινού με τις αρχές της Γεωργίας το γεωργιανό οργανωμένο έγκλημα το οποίο ε, ελέγχεται από ε, κλέφτες ε, οι οποίοι είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία της περιοχής της Βρασίας και οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε τομείς όπως είναι το τράφικινγκ, οι δολοφονίες, οι κλοπές ε, και αυτή τη στιγμή πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίσουν σοβαρά ε, προβλήματα από την εγκληματικότητα που προκαλούν αυτές οι ομάδες, ε, το, ε, η φύση αυτού του, ε, αυτών των εγκληματικών πράξεων είναι ιδιαίτερα διεθνής και γι' αυτό το λόγο είναι, πρόκειται για έναν τομέα που θα θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τους συναδέλφους μας στη Γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ πολύ και τους δύο και από τα μέλη κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο της Ευρωπόλ για την παρουσίαση αυτών των συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας. Θα σταθώ περισσότερο στη συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ευρωπόλ που είναι μια συμφωνία κλειδί που θα ενισχύσει την ε, ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύοντας αυτήν την πιο κοντινού μας γείτονα. Επίσης ε, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ σημαντική για την, ε, την αντιτρομοκρατική δράση και επίσης είναι πολύ σημαντικές οι ανταλλαγές σε θέματα πληροφοριών, αναλύσεων και πρόληψης εγκλημάτων. Καθώς είμαι ε, εισηγήτρια για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων ανάμεσα στην Ένωση και την Ουκρανία, χαίρομαι που φτάνουμε στην τελική φάση για την ολοκλήρωση αυτή τη συμφωνίας, που έρχεται να ενισχύσει το πρόγραμμα δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και στόχο έχει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει αυτή η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή για να καρποφορήσει όσο γίνεται πιο σύντομα. Θέλω δύο ερωτήσεις ωστόσο να θέσω. Πρώτον, στην επιχειρησιακή διάσταση. Μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα εγγυημένα δημοσιονομικά μέσα για την εφαρμογή της συμφωνίας, ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος και τα κονδύλια που χρειάζονται έχουν ε, προβλεφθεί ώστε οι αρχές να μπορέσουν να το περιλάβουν στον προπολογισμό του 2017 και στην ε, στρατηγική διάσταση είδαμε κάποιες ε, ε, μνήες απάντησης αλλά ακριβώς πώς θα συμπεριληφθεί αυτή η συμφωνία και πώς θα χρησιμοποιηθεί για να σημάνει προσέγγιση της στρατηγικής της Ένωσης της Ουκρανίας και της Γεωργίας για τρομοκρατική δράση, κατά πολέμηση εμπορίου ανθρώπων ή ακόμα ξέπλυμα χρήματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάμπριλ. Ο κύριο Πίτρο, μετά δεν θα ακούσουμε άλλον ε, συνάδελφο γιατί έχουμε τι ψηφοφορίε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Γεροπόλ για την εργασία τη και για τη συμβολή τη αυτή του πολύ σημαντικού οργανισμού στην ε, ενίσχυση της ε, ασφάλειάς μας και της ε, καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος στην ε, Ευρώπη. Θέλω όμως να τον σημειώσω ένα πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθεί. Το νέο κανονισμό της Europol αρχίζει να ισχύει τον επόμενο χρόνο και δίνει στο Κοινοβούλιο ένα κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο νέων επιχειρησιακών συμφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπόλ και τρίτες χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι ε, σχετικό λόγω της πολιτικής κατάστασης και την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες αυτές χώρες. Εμείς ε, ενημερωνόμαστε για τόσες νέες ε, συμφωνίες συνεργασίας τόσο λίγο χρόνο πριν από την έναρξη ισχύω νέα, της νέας συμφωνίας, της, την ανάληψη των νέων μας αρμοδιοτήτων. Βασική μου ερώτημα είναι γιατί τόσο τρέχουμε, δεν καταλαβαίνουμε που είναι, το, γιατί είναι τόσο επίγον και αν είναι δυνατόν θέλουμε να έχουμε απάντηση σε αυτή την πολύ βασική ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά με την Europol και το Συμβούλιο για όλα αυτά, αλλά παρακαλώ Α σεβαστούμε τα αποτελέσματα των τριμερών συζητήσεων που είχαμε που θεσπίζουν νέο κανονισμό και εξασφαλίζουν νέο, νέα ανοιχτή διαδικασία ελέγχου για τις μελλοντικές συμφωνίες. Επανέρχομαι στη βασική με ερώτηση. Γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ, Πρόεδρε. Um, Ευχαριστώ κύριε Πίτερσον. Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό. Είναι πολύ βασική ερώτηση. Όπως επίσης τα ερωτήματα της κυρίας Γκαμπρίαλ είναι σημαντικά. Πανέρχομαι στη Προεδρία και στη Γιουροπόλα. Παρακαλώ να μας απαντήσετε. Θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφο για το Europol, γιατί αυτό το ερώτημα είναι πιο επιχειρησιακό και ίσως μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα. Thank you, Chairman. Ε, ε, as the... Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, θα ήθελα ε, να αναφέρω τους πόρους για την εφαρμογή στόχος ε, είναι ε, να ξεμπλοκάρουν ε, το κανάλι ανταλλαγής πληροφοριών. Τα χρήματα τα οποία χρεαπαιτούνται θα σχετίζονται στη συνέχεια εν μέρη για τη δημιουργία ασφαλών γραμμών επικοινωνίας και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για υλικά γραφείου, υπολογιστές και η συνεργασία όσον αφορά αυτή τη συμφωνία που έχουμε με την Ουκρανία είναι τέτοια ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω σημαντική επένδυση όσον αφορά τη γεωργία, οι πόροι που χρειάζονται για την εφαρμογή δεν είναι τόσο μεγάλη και σε αυτό το πλαίσιο όσον αφορά το μίσο όπως είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και το trafficking ε, είναι σημαντικά ζητήματα όσον αφορά ε, το ε, ζήτημα του κόστους είναι ένα πολιτικό ερώτημα πολλές φορές συμμετείχα στις συζητήσεις για τον κανονισμό της Ιδροπόλ και θα ήθελα να υπενθυμίσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι φυσικά ο νέος κανονισμός δίνει ε, περισσότερες δυνατότητες ελέγχου στο Κοινοβούλιο, αφαιρεί όμως ε, τη δυνατότητα για την Ευρωπόλ να ε, προβεί σε σημαντικές διεθνείς ε, συμφωνίες με μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα οποία ε, στη συνέχεια γίνονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κομισιόν. Χάνουμε λοιπόν ένα κομμάτι της επιχειρησιακής μας δυνατότητας. Αυτός όμως δεν είναι ο λόγος για τον οποίο έχετε μπροστά σας τρεις συμφωνίες σήμερα. Ο λόγος είναι ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται εδώ και καιρό και πλέον έχει έρθει η ώρα να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία που ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής, ε, κράτησε περί τα δύο χρόνια και είναι και είμαστε στους τελευταίους μήνες μέσα στους οποίους νομίμως μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να σας απαντώ λοιπόν το ερώτημα. Νομίζω ότι απαντήσατε ε, τα ερωτήματα. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή τη συζήτηση όταν η κυρία Γκάμπριελ παρουσιάσει την έκθεσή της, διότι απαντήθηκαν κάποια βασικά ερωτήματα. Όταν λοιπόν παρουσιάσει την έκθεσή της θα συνεχίσουμε αυτό ε, το σημείο κλειδί για τη δική μας Επιτροπή. Επειδή Ευχαριστούμε λοιπόν για τις απαντήσεις που δώσατε. Αγαπητοί συνέδελφοι, θα συνεχίσουμε αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε θα επανέλθει η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Τώρα στις 5.40 ε, θα έχουμε μια ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν άλλο ένα λεπτό. colleagues, we just have two simple votes, so if you don't have your card... Έχουμε δύο ψηφοφορίες. Αν λοιπόν δεν έχετε μαζί σας ε, την κάρτα σας, ε, τότε μπορείτε να ψηφίσετε διαχειρός. Παρακαλώ καθίστε. Κύριε Κοέλιο, πάντοτε είστε έτοιμος εσείς, όμως δεν είναι όλοι. Including many of your colleagues, if you would like to look to your uh, left. Μαζί με εσάς όμως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, αν κοιτάξετε προς αριστερά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν είστε έτοιμοι, σε περίπτωση που δεν έχετε τις κάρτες σας, μπορείτε να ψηφίσετε διαχειρός. Ε, μπορεί κάποιος άλλος να δείξει αν έχει μαζί του την κάρτα του, η κυρία Γκάμπριελ. Πραγματικά εσείς. Ελπίζω να μην είχα πει τίποτα. Μπορείτε λοιπόν συμβούλικα να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας. Ο κύριο Κένκε και η κυρία Γκάμπριελ λοιπόν θα ψηφίσουν διαχειρός. Κάποιος άλλος εκ των συναδέλφων. Ωραία, ας περάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία που αφορά την πρόταση ψηφίσματος ε, σχετικά με την έγκριση της σύναψης ε, από την Ευρωπόλ της Συμφωνίας για τη Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Ασφάλειας της Κίνας και της Ευρωπόλ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Υιοθετείται με 30 ψήφους υπέρ, 6 κατά, 5 αποχές. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εαυτό μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ πριν. Όσον αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών, η υπήκοη των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και ε, τρίτον χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Αφορά την Ουκρανία, η συγκέντρια είναι η κυρία Γκάμπριελ και πάλι ξεκινάει η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε Τώρα στην δεύτερη τροπολογία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτη τροπολογία, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας απορριπτεται Έβδομη τροπολογία. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 4. Λήξη. Απορρίπτεται. Πέμπτη τροπολογία. Έναρξη. Λύση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Έναρξη της ε, ψηφοφορίας για το τροποποιημένο κείμενο. Λήξη. εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Και έχουμε την ψηφοφορία για τις ε, διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις ε, και τη σύνθεση της ομάδας των διαπραγματευτών. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. 38 υπέρ εγκρίνεται 5 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Και αναφέρεται η λίστα των διαπραγματευτών. Ευχαριστώ ε, τους εισηγητές αλλά και ε, τους καλεσμένους μας που βρίσκονται στην αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Και μεταξύ αυτών ε, και η αποστολή από την Ουκρανία. Η κυρία Γκάμπριελ θέλει να πει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο να πω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη στήριξή τους. Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα υποστήριξης προς το λαό της Ουκρανίας, προς τις αρχές της Ουκρανίας, όσον αφορά την εταιρική μας σχέση και πραγματικά θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς το Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν πριν αρχίσουν οι διαθεσμικές ε, αυτές διαπραγματεύσεις να τοποθετηθεί. Thank Ευχαριστώ κυρία Γκάμπριελ. Ελπίζω να εισακουστείτε από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ όλους. Sorry, colleagues, I have to do point 12, which is any other business. No. Θα πρέπει να κάνω και το 12ο σημείο, ε, διάφορα όχι, οπότε η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 29 Σεπτεμβρίου και εδώ λίγη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ.